So, dear colleagues, start? Good afternoon, everybody. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Χούμπνερ χρειάστηκε να μεταβεί στην Πολωνία για κάποια προσωπικό τη υπόθεση, επομένως θα προεδρεύσω εγώ στη σημερινή συνεδρίαση. Να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 1 της ημερήσια διάταξης, έγκρισή τη αν συμφωνείτε με τις προτινόμενες αλλαγές. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρούμε ότι εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Ο Ισπανός Υπουργός ε, θα φτάσει ο λίγο αργοπορημένος, δηλαδή γύρω στις 3.30. Ε, Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο ε, υπαριθμών 12 με τον κύριο Ευγένη Κύριλοφ και θα σου δώσω Ευγένη αμέσως το λόγο να μας παρουσιάσεις την έκθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας δώσω μια σύνδεμη πληροφόρηση σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά τις ε, διαδικασίες τροποποίησης ε, των, του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής. Όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εδώ και πολύ καιρό και έχουν, καιρό και έχουν υπάρξει κάποιες ε, ε, επιπλοκές. Το προηγούμενο μήνα ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η σχετική τροποποιητική, ο σχετικός τροποποιητικός οργανισμός της Επιτροπής ε, και επομένως ξεκίνησε επισήμως η έκθεσή μας, η εργασία μας σχετικά με τις και σύμφωνα μάλλον με τις νέες διαδικασίες της Λισαβόνας αλλά εξακολουθεί να παραμένει και μια, μια ε, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι υπάρχει επιμονή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 50 ε, του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβολίου, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρέτζη και η Επιτροπή ε, απασχόλησης ε, θα πρέπει να συνεκπονήσουν την ε, έκθεση. Εμείς ε, βεβαίως επιμένουμε ότι θα πρέπει ηγετικό ρόλο και μοναδικό ρόλο να παίξει η δική μας Επιτροπή. Όμως την προηγούμενη εβδομάδα οι πρόεδροι των Επιτροπών δεν μπόρεσαν να λύσουν το θέμα και επομένως θα πρέπει να λυθεί το θέμα στην συνεδρίαση των Προέδρων στις 4 Φεβρουαρίου. Επομένως εξακολουθεί να παραμένει αυτή η ασάφεια. Και επομένως αφενός εκφράζεται η προθυμία για καλή συζήτηση και καλή συνεργασία, ε, αλλά από την άλλη μεριά εγώ δεν είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω οτιδήποτε περισσότερο από ένα έγγραφο προς συζήτηση. Αυτό το δεύτερο έγγραφο εργασίας λοιπόν κάνει συγκεκριμένε προτάσεις που κατά την άποψή μου θα συνεισφέρουν στην ορθή τροποποίηση του περιεχομένου ε, του ε, εγγράφου. Βεβαίω, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να επιταχυνθεί η εργασία στο Κοινοβούλιο, η οποία έχει μπλοκαριστεί όπως γνωρίζετε ε, λόγω τη της αργοπορία αργοπορίας από πλευρά του Συμβουλίου. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο, ε, χωρίς καμία περαιτέρω εργοπορία, θα προχωρήσει στο θέμα της απλούστευσης και τροποποίησης ε, των ε, λόγω ταμείων. Ήδη είχα συνάντηση με συναδέλφους από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, με τους κοιόδης εισηγητής, τους εισηγητές τους ε, και νομίζω ότι τα πάμε αρκετά καλά. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο, ε, το περιεχόμενο της προτάσεως της Επιτροπής, ε, Βεβαίω ε, ε, εμείς μπορούμε να στηρίξουμε όλες τις προτάσει απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι είναι τα θέματα της χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης ε, και η επάρκεια ενεργειακών πόρων. Ε, όσον αφορά δε το εύρος ε, και το πεδίο εφαρμογής ε, και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά βεβαίως εμείς θα θέλαμε να υπάρχει η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μειωθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί από την Όλαφ. Επανειλημμένα βεβαίως εμείς και σαν Επιτροπή αλλά και σαν Κοινοβούλιο έχουμε θίξει τα θέματα αυτά και έχουμε πει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να να απλουστευθούν, να οι κανόνες και οι διεργασίες οι οποίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά ε, που ε, περιμένουμε. Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της προτάσεως της Επιτροπής θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, την οικονομική και πιστοτική κρίση που πρότεινε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα οποία συμφώνησε το Συμβούλιο ε, θεωρώ ότι δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές από το έγγραφο ε, του Ιουλίου. Εγώ προτείνω να μην αποδεχθούμε το, το, σημείο 77 όσον αφορά το κοινωνικό, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, καθώς ε, επίσης και οποιαδήποτε αναφορά για τον προπολογισμό 9-10. Ξέρετε ότι οι περισσότερες χώρες ήταν κατά των σημείων αυτών. Αντί ε, να τροποποιήσουμε το άρθρο 77, εγώ προτείνω να τροποποιήσουμε το άρθρο 82, ε, το οποίο επιτρέπει στα κράτη τα οποία έχουν περισσότερο θυγή από την κρίση να πάρουν ε, μία προκαταβολή της τάξης του 2% όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Αυτό βεβαίως αφορά λίγες χώρες αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη για τι χώρε οι οποίε έχουν ιδιαίτερο πληγή όσον αφορά το 93. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, δούμε κάποια ευελιξία όσον αφορά τι δεσμεύσεις τι ε, ε, του 2007 και πιστεύουμε ότι στι δεσμεύσει του προπολογισμού από το 2008 μέχρι το 2013 αυτή η τροποποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό ε, οι χώρες δεν θα χάσουν και τους πόρους του 2007. Ε, και αυτό νομίζω ότι αφορά μεγάλο αριθμό χωρών, τις περισσότερες χώρες και νομίζω ότι όλες θα καλωσορίσουν την ε, τροποποίηση αυτή. Γνωρίζουμε όλοι ότι το 2007 ήταν πάρα πολύ δύσκολο από των βαριών διεργασιών των λόγω προγραμμάτων. Τώρα, στο τελικά θα ήθελα να πω ότι περιμένω ότι η περαιτέρω συζήτηση θα βασίζεται σε ε, κανονικό έγγραφο εργασίας και επομένως ότι θα είναι πιο επικοδομητική η εργασία μας. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους συναδέλφους να υποβάλουν τις ε, απόψει του έτσι ώστε να έχω έτοιμο το επόμενο έγγραφο εργασίας για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ κύριε Σιγητά. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στους συντονιστές πρώτα. <clears throat> Κάποιες αποσαφηνήσεις ε, όσον αφορά το έγγραφο αυτό και όσον αφορά τον κανονισμό στο σύνολό του. Ενδεχομένως ε, δεν έχω καλή πληροφόρηση και επομένως να λαθεύω, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται ε, όσον αφορά τις γενικές διαδικασίες, γιατί από όσο ξέρω Πρώτα είχαμε την πρόταση της Κομισιόν μετά του Συμβουλίου, μετά είχαμε ε, αλλαγή των συνθήκων από την Νίκαια στη Λισαβόνα, τώρα δουλεύουμε βάσει της Λισαβόνας, αν δεν κάνω λάθος πάντα, και επομένως τώρα μόλις μπήκαμε στη συναπόφαση. Οι τροπολογίες σας αφορούν το αρχικό κείμενο της Επιτροπής ή αφορούν και βασίζονται στην συμφωνία που έγινε τον Νοέμβριο με το Συμβούλιο. Ας πούμε, το αυτό το 100% το, το περίφημο. Και για να ξεκαθαρίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Θέλω να ξέρω δηλαδή ε, ε, επί ποιου βασίζουμε την εργασία μας ε, και πώς θα προχωρήσουμε και με ποια διαδικασία θα προχωρήσουμε. Συγγνώμη για τις απλοϊκές ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω η παρουσίαση να γίνεται έτσι ώστε να είναι παρακολουθήσιμη, να μην έχει τόσο πυκνό περιεχόμενο, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τους διερμηνείς οι οποίοι πρέπει και αυτοί να μπορούν να παρακολουθήσουν για να μας εξηγήσουν επέτειλως πρόκειται. Μπορούμε να έχουμε ένα κείμενο εγγράφω αν θέλει ο μιλητής, και να αναδειφίσουμε το γραπτό κείμενο στη συνέχεια. Δεύτερον, σε όλη αυτή τη διαδικασία παρουσιάσεων υπήρξε κάτι το οποίο δεν ήταν ε, ιδιαίτερα σαφές. Εγώ κατανόησα μόναχα εκ των υστέρων, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τις διάφορες υπηρεσίες και κάναμε έλεγχο του τι συνέβη σε σχέση με τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι εμείς εργαζόμαστε από τη βάση του κειμένου της Κομισιόν από τον Ιούλιο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα πρέπει οι σκέψεις και οι προτάσεις να έρθουν σχετικά γρήγορα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τις προτάσεις μας από το Συμβούλιο, αλλά συνήθω αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το Συμβούλιο δεν λαμβάνει υπόψη τι δικέ μα προτάσει. Θα πρέπει λοιπόν και το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τι καλέ προτάσει που μπορεί να υποβάλει το Κοινοβούλιο. Επομένως δεν πρέπει να καθυστερήσει η διαδικασία, οπωσδήποτε όχι από τη δική μας πλευρά. Σας λέω και πάλι, η βασική μας εκκίνηση η βασική μας αφετηρία είναι το κείμενο της Κομισιόν και εγώ πιστεύω ότι αντί για έγγραφο εργασία θα μπορούσαμε να έχουμε μια έκθεση. Δεν έχει νόημα να παραμένουμε μόνο σε επίπεδο εγγράφων εργασία. Τα έγγραφα εργασία δεν συνοδεύονται από μια διαδικασία. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να θέσουμε τροπολογίε. Χρειαζόμαστε μια πλήρη κανονική έκθεση για να υποβάλουμε τροπολογίες. Και σας λέω και πάλι από πλευράς περιεχομένου δεν έχει νόημα να συζητάμε τη στιγμή που δεν έχουμε φτάσει στο στάδιο μιας έκθεσης. Απλώς καθυστερούμε τη διαδικασία, χρονοτριβούμε και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου να είναι το Κοινοβούλιο αυτό το οποίο καθυστερεί τη διαδικασία. Επομένως, εγώ θα ήθελα όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη συνταχθεί να τύχουν επεξεργασίας ώστε το ταχύτερο δυνατό να καταλήξουν να αποτελέσουν μια έκθεση. Για μένα δεν είναι πρόβλημα το να είναι σε λίγες γλώσσες μονάχα αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι έτοιμοι να το δεχτούν και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Μετά πρέπει να υπάρξει μια προθεσμία για τις τροπολογίες και μετά μπορούμε να κάνουμε τις συζητήσεις για το περιεχόμενο. Και έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε διατυπώσει προς τον εισηγητή εδώ και τρεις μήνες για το πού θα θέλαμε να καταθέσουμε τροπολογίες στο έγγραφο της Κομισιόν. Και είμαστε έτοιμοι να τα διατυπώσουμε αυτά και σε γραπτή μορφή. Απλώς πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο βάση και να υπάρχει μια κείμενη διαδικασία. Γι' αυτό εγώ προτείνω το ταχύτερο δυνατό να εκπονηθεί μια έκθεση από την πλευρά του εισηγητή. Είναι γεγονός ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στο έγγραφο της προηγούμενης Κομισιόν, ό,τι και να συμβεί. Αν υπάρχει μεγάλος βαθμός σύμπνοιας με το Συμβούλιο, θα πρέπει ο συγητής να αντιδράσει με τον τρόπο αυτό, με τις τροπολογίες του και να προσεγγίσει τη θέση του Συμβουλίου. Και σίγουρα χρειαζόμαστε μία προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών σε ένα επίσημο έγγραφο το οποίο είναι έκθεση και μόνο τότε μπορούμε να περάσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία και σας ζητώ αυτή η διαδικασία να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό και όχι να έχουμε συνέχεια καθυστερήσεις. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Βανίστερόι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε σχετικά με την ερώτηση που έθεσε ο Στάνος προηγουμένως σχετικά όσον αφορά αυτό το καθεστώς δηλαδή του εγγράφου εργασίας. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι ε, πραγματικά ο εισηγητής θα πρέπει να μας πει τι θέλει. Ε, γιατί αν πρέπει να δεχτούμε τη δέσμη θα πρέπει να ξέρουμε με τι συμφωνούμε. Βεβαίως μπορούμε να δούμε τις επιθυμίες, των, τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου και να τις υποβάλλουμε, ε, γνωρίζοντας πάντως ότι θα πρέπει να εργαστούμε με κάποια σχετική ταχύτητα, ε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και επομένως ε, να θεωρήσουμε ότι όλα πάνε προς την καλή κατεύθυνση και επομένως τότε να μπορέσουμε να πάρουμε θέση όσον αφορά τις τροπολογίες. Επομένως, θα ήθελα να μας πει ο εισηγητής εάν θα μας προτείνει να ακολουθήσουμε την διαδικασία ε, όπως θέλουμε εμείς, ε, με το δικό μας αριθμό ή εάν θα ακολουθήσουμε την θέση του Συμβουλίου, δηλαδή όσο πιο γρήγορα, να ε, πάρουμε απόφαση και να μας πει και η Επιτροπή επίσης τη θέση της. Ευχαριστώ. Ο ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να κάνουμε αυτή την ε, απλοποίηση ε, των απαιτήσεων κάποιων ταμείων. Όμως θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά όσον αφορά ας πούμε τα μεγάλα περιβαλλοντικά στοιχεία, ε, ε, ε προγράμματα. Στα μεγάλα ε, λοιπόν προγράμματα δεν νομίζω ότι ε, θα τους κάνει καλό να τα μειώσουμε και νομίζω ότι το όριο των 25 εκατομμυρίων ήταν πάρα πολύ καλό γιατί τα μεγάλα προγράμματα δεν είναι απαραίτητα τα καλύτερα. Επομένως το να πούμε ότι ε, θα χρηματοδοτήσουμε από 50 εκατομμύρια και πάνω δεν με βρίσκει πολύ το σύμφωνο και τα μικρά προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Mr. Ε, Goodmanis. please. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Έχουμε δύο θέσεις εδώ. Έχουμε δύο θέσεις εδώ, είπα. Η μία είναι του Συμβουλίου, η οποία φυσικά ακολουθεί την θέση της Κομισιόν. Το πιο ενδιαφέρον είναι να θέσουμε το εξή ερώτημα στον εισηγητή. Στις δικές του προτάσεις, στις δικές του τροπολογίες, αυτός ο ίδιος στην τροπολογία, μια στιγμή να βρω τα χάτια μου, στην τροπολογία υπαριθμών 11, στο έγγραφο εργασίας του, ο εισηγητής, λέει ζητάει τη διαγραφή του κειμένου της Κομισιόν στο σημείο αυτό. Από ό,τι κατανοώ, η διαφορά μεταξύ της θέσης της Κομισιόν και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση και τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση στο Κοινωνικό Ταμείο γιατί αυτό λέει η Κομισιόν, όταν ζητείτε πληρωμή στα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 100% το 2009 και το 2010, Αν υπάρξει λοιπόν μια τέτοια απόφαση, η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί με συναπόφαση. Δεν είναι στο χέρι του Συμβουλίου να αποφασίσει. Σας λέει λοιπόν το Συμβούλιο ότι η αρχή αυτή του 100% χρηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν τα κράτη-μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι όλες αυτές οι πληρωμές αδειρήτως απαιτούνται ως μέτρα αντιπολε... αντιμετώπισης της κρίσης. Επομένως, δεν πρόκειται για τον αριθμό των χωρών που έχουν επικαλεστεί ιδιαίτερες συνθήκες για να έχουν μεγαλύτερες πληρωμές. Το Συμβούλιο λοιπόν κάνει μια πρόταση η οποία τροποποιεί την πρόταση της Κομισιόν προς τα κάτω, προς τα ίσονα. Αν θέλει κανείς λοιπόν να επιτύχει το 100% της πληρωμής από την Κομισιόν, θα πρέπει να καταδείξετε ότι πρόκειται για μέτρα αντιπροτόψης της κρίσης, τα οποία μέσω του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσετε το 2009 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2002 και εσείς στις τροπολογίες σας. Ζητάτε να ακυρωθεί, να διαγραφεί η πρόταση της Κομισιόν. Και ρωτώ. Επομένως, εσείς προτείνετε αυτό το υποστηρίζετε αυτό που λέει το Συμβούλιο ή όχι στο έγγραφο εργασία. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Τα άλλα είναι απλώς διαδικαστικά και τυπικά και τυπολατρικά αν συμφωνούμε με εσά στις τροπολογίες σας, τότε δεχόμαστε θέση του Συμβουλίου. Ότι δηλαδή το... η Κομισιόν μπορεί να πληρώσει για το Κοινωνικό Ταμείο για τα έτη 2009 και 2010 100% με την προϋπόθεση ότι το κάτω μέλος θα αποδείξει ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για μέτρα κατά της κρίσης. Για μένα δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό γιατί όλοι θα πούνε για την κρίση τα θέλουμε τα λεφτά. Γι' αυτό αυτό είναι ένα θέμα όπου θα ήθελα πραγματικά να έχω την άποψη του εισηγητή. Αυτό ήταν και θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Όρη. Αλλά η πρότασή σας, η θέση σας στην τροπολογία 11 είναι να αντικαταστήσετε την πρόσθεση της Κομισιόν με τι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, σε πέντε λεπτά αν είναι δυνατόν να απαντήσετε, διότι ο Ισπανός Υπουργός είναι καθοδόν, αλλιώς θα συνεχίσουμε μετά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, εγώ λυπάμαι που ίσως διάβασα πάρα πολύ γρήγορα το κείμενο, ε, αγγλικά ήταν πιο εύκολο να το καταλάβουν όλοι, γιατί έτσι κι αλλιώς μισή ώρα έχουμε εδώ πέρα. Αλλά το τόνισα και έτσι κι αλλιώς θα στείλω σε όλους τους συναδέλφους την ομιλία μου, Περί τίνο πρόκειται. Τώρα βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι είναι το πιο σημαντικό να καταλάβουμε. Εγώ δεν έκανα τίποτα το εφάνταστο ή το δημιουργικό. Πήρα το κείμενο της Κομισιόν και προσπάθησα να δω τι έχει προκύψει μετά τις συζητήσεις του Συμβουλίου και πώς να αντανακλώνται αυτές οι τροπολογίες μετά από τις συζητήσεις του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο θέλω να δω λοιπόν είναι πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Με ρωτάτε, αλλά και εγώ σας ρωτάω. Πώς πάμε προς τα μπροστά. Πάμε. Προχωράμε με ταχύτητα για να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να, το, να θεσπίσουμε αυτή την αρχή ώστε να λειτουργήσει από τον Απρίλιο ή θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τη φυσιολογική διαδικασία στην απόφαση. Δεν υπάρχει καμία φαντασία η οποία εμπλέκεται. Γιατί αυτό είναι το τροποποιημένο έγγραφο της Κομισιόν μετά από τη Λευκή Βίβλο. Λυπάμαι κυρία Σρέντερ. Το Κοινοβούλιο δεν φταίει καθόλου. Γιατί περιμένουμε συνέχεια για το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε ότι φταίμε. Και το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή Απασχόληση θέλει και αυτή να έχει μια συνεισυγεσία για το θέμα αυτό. Και γι' αυτό μιλάμε ακόμα για επίπεδο εγγράφου εργασία. Γιατί εναπόκειται στη συνέλευση των Πρόεδρων να αποφασίσει αν εμεί είμαστε η επί τη αρχή επιτροπή για το θέμα αυτό ή όχι. Και ακόμα συνεχίζουμε να περιμένουμε και γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Επίση. σε ό,τι αφορά την τροπολογία υπαριθμών 11, που Τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Όπως ξέρετε η αρχική πρόταση ήταν του, της Κομισιόν, έχει διαγραφεί. Τώρα η νέα πρόταση αφορά μονάχα τις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο. Και εδώ αναφέρεται ότι οι χώρες αυτές είναι, <coughs> είχαν μείωση του ΑΕΠ το 2009 σε σχέση με το 2008 10% σε πραγματικούς όρους. Ε, πόσες θα είναι, δύο-τρεις χώρες θα είναι. Οι υπόλοιπες χώρε προφανώ δεν μπορούν να υποφεληθούν από τέτοια μέτρα. Και υπήρχε μονάχα ένα σχόλιο για τα 25 ή 50 εκατομμύρια για τα μεγάλα σχέδια. Αρχικά το είχε προτείνει η Κομισιόν για να μην υπάρξει διαφορετική μεταχείριση γιατί κάποια κράτη-μέλη διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά αυτό θα το δείτε όταν έχουμε ήδη ένα έγγραφο εργασία και να δούμε ποια είναι η γενική άποψη που επικρατεί. Αυτά μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι στις 22 Φεβρουαρίου θα υποβληθεί το προσχέδιο προς έγκριση. Okay. Καλωσορίσατε λοιπόν κύριε Υπουργέ. Σας καλωσορίζω εξ ονόματος ολόκληρης επιτροπής. Ο κύριος ε, Κάρλος ε, Οκάνια, Υφυπουργός Οικονομικός, Οικονομικών, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, θα μας ε, κάνει μια παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή. Έχετε τον λόγο κύριε Υπουργέ. Κυρίε και κύριοι, βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας αναλύσω την παρούσα κατάσταση της περιφερειακής πολιτικής και να σας παρουσιάσω και τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στο θέμα αυτό θα αναφερθώ σε τρία στοιχεία τα οποία θεωρώ κλειδί για την ε, περιφερειακή πολιτική, που είναι το μέλλον της πολιτικής συνεχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ολοκλήρωση της ε, αρχής της ε, εδαφικής συνοχής και η απλούστευση της νομοθεσίας της πολιτικής συνοχής. Όπως είναι λογικό, αυτά τα τρία θέματα θα αναλυθούν εις βάθος στη διάρκεια του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας και θα περάσω τώρα στην διεξοδικότερη ανάλυση τους θα σταθώ καταρχάς στο μέλλον της πολιτικής συνοχής. Στη διάρκεια του εξαμήνου και υποθέτω και στα μελλοντικά εξάμεινα, το μέλλον της πολιτικής συνοχής θα αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο ανάλυσης και συζήτησης, τόσο από πλευράς ε, ε, προοπτικής, ε, των καθορισμού των προτεραιοτήτων, όσο και των στόχων. Η, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βιώνει την πιο σημαντική οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών και αυτό κατέδειξε το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλές χώρες και περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο επίπεδο ε, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και θα υπάρχουν επιπτώσεις όταν θα δούμε την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης ε, ανάπτυξη συγκεκριμένων διαρθρωτικών αλλαγών που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη και στις ε, περιφέρειες να οργανωθούν καλύτερα και να λάβουν υπόψη τους τις αένας αλλαγές που έχουν γύρω τους και να κάνουν και μακροπρόθεσμες αλλαγές. Δεύτερον, η κρίση κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε και να προβλέπουμε μηχανισμούς ευέλικτους ε, απάντησης ε, βραχυπρόθεσμα σε οξύες περιπτώσεις κρίσεως όπως ε, την πρόσφατη, σοκ τα οποία δυστυχώς πολύ δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε και που πλήττουν τις περιφέρειες σε πολύ σημαντικό βαθμό, ασύμετρα θα λέγαμε. Η δυνατότητα λοιπόν οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών αυξηθούν στο εγγύς μέλλον είναι καθόλου υπαρκτή και είναι πολύ πιθανό στα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια επιβράδυνση της διαδικασίας, της διαδικασίας σύγκλησης ε, μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, στην ε, μικρότερη οικονομική ανάπτυξη, με μικρότερε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και μεγαλύτερο περιορισμό στον ε, προπολογισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση ε, την οποία θα μπορέσουν κάποιες άλλες περιοχές να τις εκμεταλλευτούν και κάποιες άλλες όχι και να μείνουν ακόμα πιο πίσω από τις η οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα οικονομία κοινωνική που θα είναι πιο βιώσιμη, θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και θα είναι πιο καινοτόμα. Και επίση η κρίση είναι μια ευκαιρία για να αναδιαθρώσουμε την πολιτική μα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο βιώσιμο μέσο. Όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές οι συνιστώσεις της κρίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, η οποία αδιαφυσβήτητα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, ε, πολύ ισορροπημένη ένταξη των διαφόρων περιορισμών και τις ε, ίσες συνθήκες εντός των περιφερειών. Οι φάσει τη οικονομική επιβράδυνση, ε, τουλάχιστον στο παρελθόν, είχαν αρνητικέ επιπτώσει στη σύγκληση. Ε, οι, πιο, λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές συνήθως είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και ίσως ε, μπορεί να συμβαίνει αυτό γιατί δεν υπάρχουν πιο συμπαγείς δομές για να το στηρίξουν. Στα πλαίσια αυτό λοιπόν η ε, περιφερειακή ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει να μετριαστούν οι επιπτώσεις. Η Ευρώπη είναι υπέρ της σύγκλησης και το κάνει αυτό γιατί είναι το ε, βασικό στοιχείο σταθερότητας ε, τόσο πολιτικής όσο και νομικής για τις περισσότερες χώρες μέλη. Αλλά και γιατί η ενιαία αγορά το να γνωρίζει κανείς καλύτερα τους πολίτες των διαφόρων κρατών μελών και να γνωρίζει καλύτερα τους κανόνες και τους εθνικούς θεσμούς δίνουν καλύτερες δυνατότητες για μια οικονομία αγοράς. Η πολιτική συνοχή ε, συνεισφέρει στην ολοκλήρωση, στην ε, αλληλεγγύη και στη συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σύγκληση στι ε, λιγότερο εύπορε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πολιτική συνοχή θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι παρούσα σε όλη την έκτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 είναι αδιά, αναπόσπαστο στοιχείο στο σχεδιασμό των μελλοντικών κοινοτικών πολιτικών και είναι κάτι το οποίο να απαραίτητο στα επόμενα δέκα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης οικονομικής που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και θα είναι πιο κοινωνικά ε, σωστό. Η πολιτική συνοχή συνεισφέρει ε, στις πολιτικές οικονομικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο κλειδί στο σχεδιασμό της στρατηγικής του 2020 όπως είναι και για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Χωρίς να ξεχνάμε λοιπόν τις επενδύσεις και σε υποδομές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη σε πολλά κράτη-μέλη, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες θα ε, πρέπει να διαδραματίζουν ένα όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ε, πολιτική αυτή, χωρίς να ξεχνάμε επίσης και τις ψυχευτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η ανάγκη να επαναπροσανατολίσουμε τις δαπάνες ε, για τη στρατηγική του 2020 ε, καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ε, δεν πρόκειται μόνο για κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό διότι πολλά από τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας διαπιστώνονται ότι είναι στα χέρια των περιφερειών. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία λοιπόν που δίνουν ένα επιπρόσθετο όφελος στην ε, περιφερειακή κοινοτική πολιτική είναι το γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αυτή την τεχνογνωσία θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει επίση ε, να λάβουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό τη πολιτική συνοχή και τον καθορισμό των στόχων τη. Όσον αφορά το στόχο τη σύγκληση, φαίνεται να υπάρχει μια ε, γενική συνένεση για τη συνέχειά τη και επίση θα πρέπει να αναλώσουμε και τη δυνατότητα να εισαγάγουμε και κάποιε τροποποίησει που θα τον ενισχύσουν και θα τον κάνουν πιο αποτελεσματικό. Ε, μία σημαντική πτυχή την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ είναι ο στόχος λοιπόν της σύγκλησης. Αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες χρηματοδότησης είναι ευρύτατες μέσω του ΦΕΝΤΕΡ και ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε μια αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, ε, όταν υπάρχουν νέες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα οι κλιματικές αναγές, η μετανάστευση ή η δημογραφική πίεση, θα πρέπει να υπάρχουν ε, και νέοι τομείς δράσης ε, και θα πρέπει να αναλύσουμε αφενός ε, εάν η πολιτική της νεχής αποτελεί το χρήσιμο μέσο, και αν είναι αποτελεσματική για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αφετέρου πώς θα πρέπει να διαρθρωθεί για να τις αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ε, ο περιορισμός του προϋπολογισμού είναι όλο και περισσότερος και στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο σημαντικός για πολύ μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Και ε, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες, ε, οι πόροι θα είναι όλο και λιγότεροι, γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να έχουμε και μια σειρά από δράσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ευρείες για να μπορέσουν να λάβουν υπόψη τις ιδιωτηρότητες κάθε περιοχής και τα προβλήματα σύγκλησης που έχουν. Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή είναι να καθορίσουμε τις μεταβατικές περιόδους για τις ε, περιοχές οι οποίες βγαίνουν από το στόχο της σύγκλησης. Είναι πολύ ε, λογικό να αυξηθεί ο αριθμός ε, των περιπτώσεων αυτών στο μελλοντική περίοδο προγραμματισμού και επίσης για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη στις περιοχές αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν στρατηγικές για να ε, βγούμε από, την, ε, το στόχο της σύγκλησης ε, και ο στόχος θα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν απότομες αλλαγές και να υπάρχει και μια κάποια οικονομική σταθερότητα στη διάρκεια εξόδου. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για την περίοδο προγραμματισμού που συζητάμε τώρα, Υπήρξαν και κάποιες μεταβατικές περίοδες ε, στις οποίες η χρηματοδότηση ήταν πολύ περιορισμένη και κυρίως ε, εστιάζουν στις πρώτα, στα πρώτα χρόνια της εξόδου και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ένα προγραμματισμό το οποίο θα λάβει υπόψη και την ανάπτυξη των ε, περιοχών που επηρεάζονται από το θέμα αυτό. Αυτό δημιούργησε πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές που είναι είτε στη φάση του phasing out είτε στη φάση του phasing in. Ε, αυτό ε, θα παραμείνει και θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις για τις περιφέρειες οι οποίες θα βρίσκονται σε μεταβατικές περιόδους το διάστημα 2014-2020 και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ε, προβλήματα στη χρηματοδότησή τους. Όσον αφορά τώρα το στόχο της ε, περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και την απασχόληση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα και επίσης θα πρέπει να θεμελιώσουμε καλύτερα την κοινωνία της γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση στην πρόσβαση και ταυτόχρονα να ευνοήσουμε την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού ε, και να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο των περισσότερων και καλύτερων θέσεων αποσχόληση. Στην επίμενη περίοδο προγραμματισμού τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών περιφερειών θα αποτελέσουν τμήμα αυτού του στόχου. Η στρατηγική του 2020 ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι επιλέξιμες αυτές οι περιφέρειες ε, στην πολιτική συνοχή και ίσως το προστιθέμενο όφελος, το πιο σημαντικό, να είναι ακριβώς ότι θα υπάρχει μια θετική όθηση για όλα αυτά. Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα μέσο το οποίο ε, δεν είναι μόνο ε, κατανομή πόρων αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει δυνατότητες στις διάφορες περιφέρειες, να ε, άρει αδυναμίες και να διευκολύνει διάφορες θεσμικές αλλαγές. Ε, μία άλλη πτυχή την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι στον ορίζοντα το 2014-2020 ο στόχος αυτός θα αφορά περιφέρειες ε, επίπεδου ανάπτυξης πολύ διαφορετικού και στην πραγματικότητα ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος καθορίζεται μέσω του αποκλεισμού. Μία περιοχή μπορεί να είναι ανταγωνιστική ε, εάν ε, δεν έχει σύγκληση. Αυτό σημαίνει ότι για το 2014 ο στόχος αυτός αποτελείται από περιφέρειες που, είναι, που έχουν ένα 85% εισοδήματος ε, ε, κατά κεφαλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και περιοχές που ξεπερνούν το 200% σε αυτό το μεσόρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν θα καθορίσουμε και τι δράσεις θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. Για να μειώσουμε την ε, κατανομή του κατακεφαλίου σε αυτό το στόχο, θα πρέπει να μελατώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε διάφορα στάδια. Ε, είναι πολύ λογικό σε μια περιοχή με χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα από το μέσο κοινοτικό όρο να πρέπει να βρισκόμαστε πολύ, να είμαστε μάλλον συγγνώμη, πιο κοντά σε μια περιφέρεια σύγκλησης από ότι οι ανάγκες ε, μιας ε, περιφέρειας πιο εύπορης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βασικό στόχος για τη συζήτηση είναι το, η οικονομική χρηματοδότηση. Αυτό δεν θα λυθεί με επιτυχία αν δεν καθορίσουμε σαφώς τα κριτήρια ανάθεσης των πόρων σε κάθε χώρα και κάθε περιοχή συνεργασίας ε, και επίσης τα διάφορα επίπεδα ε, ή χώρου συνεργασίας, εδαφικής συνεργασίας ε, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ε, τεράστια πλούστευση για τη διαχείριση ενός στόχου πάρα πολύ πολύπλοκου που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ε, φορέων ε, των διαφόρων χωρών που βρίσκονται και τη τερογενή φύση τους. Εάν αναλύσουμε τα διάφορα κεφάλαια του στόχου και πάλι έχουμε σημαντικά στοιχεία που αξίζουν συζήτηση. Καταρχήν σε σχέση με τη διασυνορική συνεργασία για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις προκλήσεις των περιφερειακών αυτών περιοχών και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη χρήση του δυναμικού τους. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια οριζόντια μορφή συντονισμού με όλους αυτούς τους στόχους και τις τομεακές πολιτικές. Είναι επίσης και μια καλύτερη κάθετη συντονιστική δράση γιατί η, η κατανομή είναι πολύ διαφορετική. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχύσουμε λοιπόν και την διοικητική ικανότητα για να έχουμε μια καλύτερη Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να ανακαθορίσουμε ποιοι είναι οι χώροι οι οποίοι καλύπτονται από αυτές τις ενέργειες Από την πλευρά των ευρωπαϊκών περιοχών, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιε είναι οι περιοχές οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους γιατί δεν έχει πολύ νόημα να συμμετέχει μια περιοχή σε χώρους οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους Θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη μορφή ορισμού των χώρων συνεργασία, ώστε η κάθε περιοχή να μπορεί να βρίσκεται στο φυσικό τη χώρο συνεργασία με άλλε ευρωπαϊκέ περιοχέ, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απλοποίηση. Ο ορισμό των χώρων, όπω το έχω διατυπώσει, είναι κάτι το πεπλεγμένο, αλλά θα μα βοηθήσει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε στο μέγιστο την αποτελεσματικότητα τη συνεργασία και επίση να προχωρήσουμε στο να συντάξουμε του κατάλληλου δείκτε Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία σαν στοιχείο εδαφικής συνοχής, ώστε οι περιοχές, οι ευρύτεροι χώροι και οι περιοχές συνεργασίας να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η διαμεθοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να λάμβανε υπόψη και τις αναγκαιότητες και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών αρχών και περιφερειακών και να δώσει ένα πλήρες φάσμα δράσεων. Και έρχομαι τώρα στο θέμα της εδαφικής συνοχής. Για τα θέματα του μέλλοντος λοιπόν της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ολοκλήρωση της αρχής της εδαφικής συνοχής. Η Συνήκη της Λισαβόνας έχει θέσει στο άρθρο 3 την εδαφική συνοχή ως ένα απαράγραπτο και σημαντικό στόχο για τη, σημαντική, για τη μελλοντική μάλλον πολιτική συνοχής μαζί με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Επίσης η κρίση με τις ασυμμετρικές της ε, με τους ασυμμετρικούς κλειδονισμούς έχει αυξήσει τη σημασία της εδαφικής συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δώσει νέα όθηση σε αυτή τη συζήτηση. Τον Οκτώβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πράσινο βιβλίο που είναι η απαρχή ενός ευραίος δημοσίου διαλόγου για την εδαφική ε, συνοχή σε όλες τις πολιτικές πτυχές του. Θέλει να εξασφαλίσει λοιπόν την δυνατότητα να είναι ε, βιώσιμες αυτές οι πόλεις και οι περιοχές, επίσης να υπάρχει συνεργασία μεταξύ περιοχών. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια μεγαλύτερης συνεκτικότητας των πολιτικών, ώστε να μπορέσουμε να, να συμβάλλουμε σε μια συλλογή και συμπίληση δεδομένων για όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ η πρόθεση της Ισπανικής Προεδρίας είναι να προωθήσει αυτές τις συζητήσεις και να προχωρήσει σε πρακτικές εφαρμογές αυτής της αρχής. Το τρίτο στοιχείο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι η απλοποίηση της, δι... της διαχείρισης. Αυτό είναι το τρίτο κομβικό σημείο για την ανάλυση και τη συζήτηση των εφερχόμενων μηνών. Είναι η απλοποίηση της ρύθμισης και των διαδικασιών που άπτονται της πολιτικής συνοχής στην πράξη η διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης είναι υπερβολικά απεπλεγμένη. Και αυτό οδηγεί σε μια υπερβολική και όχι δικαιολογημένη αύξηση του φόρτου εργασίας στα θέματα αυτά, κάτι το οποίο πλήττει την επιτεύξη των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, που είναι ακριβώς η στόχοι της πολιτικής συνοχής. Η τωρινή μορφή των συστημάτων ελέγχου χαρακτηρίζεται από δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα, η αύξηση της πολυπλοκότητας των ελέγχων χωρίς οι νέες αυτές απαιτήσεις να έχουν συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στο να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των κυρωτικών ταμείων. Και επίσης ό,τι αφορά την ε, διαχείριση, η διαχείριση των ε, ε, πόρων που αφορούν τα κοινωτικά ταμεία και οι επενδύσεις δεν βρίσκονται σε στενή σύνδεση. Δεν, δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε μία σύνδεση μεταξύ επίπεδου επενδύσεων και χρηματικής συνεισφοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι τα ποσά που εκταμιεύονται από τους κυρωτικούς πόρους είναι απλώς μια πολιτική μεταφοράς πιστώσεων χωρίς να επιτυγχάνουν τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε πολλούς προϋπολογισμούς για την έλλειψη πιστώσεων και ρευστότητας. Και αυτό επηρεάζει πολλούς από τους φορείς. Αναγκάζει πολλούς φορείς να προσφύγουν σε πηγές χρηματοδότησης που είναι δύσκολοι σε εποχή κρίσης και επισύρουν ένα πρόσθετο οικονομικό κόστος ιδιαίτερα υψηλό. Πολλές φορές λοιπόν δεν είναι και επιλέξιμοι αυτοί οι φορείς για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτή τη χρηματοδότηση και αυτό περιορίζει μέχρι και 10% τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των φορέων λόγω υψηλού κόστους. Σε ό,τι αφορά τα ελεκτικά συστήματα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι σαφές ότι η αύξηση πολυπλοκότητας των ελέγχων οδήγησε σε μια βελτίωση στην αποτελεσματικότητα και το ελεκτικό συνεδρίο τόνισε το 2008 την ανάγκη να λαμβάνει υπόψη η προσθέμενη αξία όλων αυτών των ελέγχων. Είναι φυσικά απαραίτητο να έχουμε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι εξασφαλίζουν το ότι είναι προσαρμοσμένοι οι πόροι οι οποίοι δίνονται στους στόχους αυτούς. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε ακεραιόφρονες του ελέγχου, χάρη του ελέγχου, κάτι που οδηγεί σε απόδοση όλο περισσότερων πόρων στον έλεγχο σε βάρος της επίτευξης των στόχων μας. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την τελευταία έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξαν ατασταλίες, μόνο σφάλματα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι ατασταλίες. Και πράγματι, παρά το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας πολλών από τα προγράμματα, το ελεκτικό συνέδριο δεν διεκρύβωσε καθόλου ατασταλίες. Ούτως ή άλλως αυτά τα σφάλματα μπορούν να προκύπτουν από μια λανθασμένη εφαρμογή των ρυθμίσεων που ιδιαίτερα πεπλεγμένες σε ό,τι αφορά την καταβολή ποσών. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει υποψία απάτηση. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να προχωρούμε στον τομέα της απλοποίησης, ώστε να καταλήξουμε σε μια διαχείριση η οποία θα είναι όσο δυνατόν πιο αυστηρή, αλλά η οποία θα εξασφαλίζει τη σωστή χρήση όλων αυτών των ποσών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή εξετάζει την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού των Διαφορετικών Πόρων. Ήδη στο τέλος του προηγούμενου έτους επιτεύχθη μια συμφωνία στο Συμβούλιο για να υπάρξει αυτή η τροποποίηση. Στην πρόταση η οποία δόθηκε στο Κοινοβούλιο υπάρχει μια σειρά μέτρων τα οποία έχουν σαν στόχο να ευκαμπτοποιήσουν τη διαχείριση χωρίς να υποσκάψουν την δημοσιονομική πειθαρχία και την αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων και του Ταμείου Συνεχής. Επομένω, <clears throat> και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη λόγω των δυσκόλων συνθηκών που περνούν τα περισσότερα κάτι σε επίπεδο προπολογισμού. Τα μέτρα αυτά δεν είναι μονάχα συγκυριακά. Είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μακροπρόθεσμα. Αλλά είναι απαραίτητο να δώσουμε έμφαση σε αυτέ τι προσαρμογέ λόγω των προβλημάτων ρευστότητα πολλών κρατών μελών. Η Κομισιόν δεν έχει προβλέψει να παρουσιάσει πρόσθετα νομοθετικά πακέτα ούτε φέτο ούτε στο υπόλοιπο τη περίοδου προγραμματισμού. Η Ισπανική Προεδρία έθεσε τον εαυτό τη ω στόχο να συνεχίσει τι εργασίε στον τομέα αυτό και αν δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αυτού του κανονισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να καθορίσουμε οδηγές γραμμές και γενικές αρχές για το σύνολο του κανονισμού των διαφορετικών ταμείων που θα έλθει ο νούπο. Στέκομαι τώρα και σε ένα θέμα το οποίο ίσως δεν βρίσκεται στον πυρήνα των αναλύσεών σας, αλλά το οποίο έχει και αυτό μια κάποια σημασία. Βάσει του άρθρου 30 του Γενικού Κανονισμού των Διαφορετικών Ταμείων, κάθε τη διάρκεια του, του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας το αργότερο τον Απρίλιο του 2010, πρώτα Απριλιά μάλιστα, η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια στρατηγική μελέτη η οποία βασίζεται στις συμβολές των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2009 με τις εκθέσεις τους. Σε αυτέ τι εκθέσει αναλύεται το επίπεδο επίτευξη των στόχων που είναι παρόντε στον προγραμματισμό των διαφορετικών ταμείων και η συμμετοχή των στόχων αυτών στου γενικότερου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο θα αναλύσει ενδελεχώ την έκθεση τη Κομισιόν και θα καταλήξει σε συμπεράσματα για αυτή την έκθεση πριν από τον Ιούνιο του 2010. Μία από τι καταστάσει που έχουν προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία του, του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συζήτηση για το μέλλον τη πολιτική συνοχή θεωρώντα ότι το εξάμεινο τη ισπανική Προεδρίας μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τη σημασία τη πολιτική συνοχή. Από αυτή την άποψη, η εξέταση τη στρατηγική έρευνα της έκθεσης θα μα επιτρέψει να καθορίσουμε καλύτερα, να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμμετοχή τη πολιτική συνοχή στις, και την θέση που πρέπει να έχει στι μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικέ. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών πολιτική. Ε, Περιφερειακής θα γίνει στη Σαραγώσα στις 19 Φεβρουαρίου και τα θέματα προτεραιότητας εκείνη τα εξής. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής που περιλαμβάνει και την εδαφική συνοχή. Η νέα προσέγγιση για τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Και τρίτον, οι κατευθυντήρες γραμμές απλοποίησης της πολιτικής συνοχής. Όπως ακόπως βλέπετε, αυτά είναι τα κύρια θέματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή επιτάπητο σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Όπω είπα και στην αρχή, περιμένω αυτό το εξάμεινο τη Ισπανική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμεύσει για να μπορέσει να δείξει την αξία τη πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τη και την σωστή τη εφαρμογή. Το έργο τη Επιτροπή σα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ισπανική Προεδρία λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχετε ήδη ε, συσσωρεύσει σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά θέματα. Η Ισπανία εξάλλου έχει μια μεγάλη πείρα και είναι ένα παράδειγμα των εξαιρετικού επίπεδου αποτελεσμάτων που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περιφερειακή πολιτική αν τα πράγματα γίνονται καλά. Αυτή η, ικανοποίηση δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να εφησυχάζουμε. Είναι πολλά κόμματα τα οποία πρέπει να γίνουν και να βελτιωθούν ακόμα και στην Ισπανία και θα συνεχίσουμε τι προσπάθειές μα προ την κατεύθυνση αυτή. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει ένα καλύτερα, ακόμα καλύτερο πλαίσιο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί περαιτέρω αυτή η πολιτική συνοχή. Θέλω λοιπόν να σα ευχαριστήσω για τη δική σα συνεργασία και να σα υποσχεθώ και ότι και η Ισπανική Προεδρία θα πράξει όλα τα απαραίτητα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας για την Περιφερειακή Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε την συζήτηση δίνοντας πρώτα τον λόγο στους συντονιστές, αν το επιθυμούν. Ο κύριος Βανίστερόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Spanje, en die zijn, zijn rijkelijk, om zo uit te drukken. γνωρίζομαι όλοι πολύ καλά την ε, εμπειρία που έχει η Ισπανία όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την ε, πολιτική συνοχή. Είναι σημαντικό ε, να ξέρουμε ότι ανέλαβε τα ενία της Ευρώπης η χώρα η οποία, στην οποία μάλλον ε, η πολιτική συνοχή έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Συνειδητοποιείται βεβαίω το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο με την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει πλέον διαφορετική θέση κυρίως όσον αφορά τις ανακοινώσεις, τις ε, ε, σχέσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να παίζουμε σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Είμαστε άρρηκτο τμήμα της διαδικασίας τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, επομένως. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Δεν ξέρω επίσης αν ε, προτίθεστε να εμπλέξετε το Κοινοβούλιο ενεργότερα στην ε, Σαραγώσα. Και να πω και το εξής. Στην αρχή της παρέμβασής σας αναφερθήκατε στρατηγική 2020 και τοποθετηθήκατε με ένα πνεύμα ε, ανοιχτό. Και εμείς το ίδιο άλλωστε λέτε περιφερειακή πολιτική, η πολιτική συνοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και βεβαίως συμφωνούμε απολύτως μαζί μας. Αλλά διαβάζοντας το κείμενο για την ορίζοντα 2020 διαπιστώνουμε ότι αυτός ο άρρηκτος κατά την άποψή μας δεσμός ε, με την, σχέση, με την συνθήκη της Λισαβόνας δεν διαφαίνεται αρκετά. Και επομένως εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε από σας ε, ότι ε, όχι έχουμε, έχετε κάποιους στόχους αλλά έχετε και συγκεκριμένα εργαλεία ε, για να προωθήσετε τους στόχους αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πόσο δεσμευμένος είσαστε σε αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα δεν θα ήταν ε, να ε, πάρουμε δύο-τρεις ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε συνολικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα. Είναι πολύ καιρό που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ξεκινήσει πράγματι τι θα πρέπει να γίνει με τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πράγματι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ισπανική Προεδρία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ισπανία τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Εγώ επίσης χαίρομαι για το γεγονός ότι αναφερθήκατε στο θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών. Και έτσι κι αλλιώς θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή διεκπεραιώνεται, αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κανονισμό ο οποίος είναι μια de παραλλαγή των ρυθμίσεων αυτών γιατί το Συμβούλιο είχε πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλήξει σε μια πιο ευρύτερη συμφωνία. Αναγκάστηκε η Κομισιόν να αποσύρει την αρχική της πρόταση και να υποβάλει μια νέα πρόταση όπως λέει και ο κύριος Φανλίστεροι. Εμείς Θέλουμε να τροποποιήσουμε αυτήν την ε, νέα πρόταση Κομισιόν με το να συνεισφέρουμε με τις δικές μας συνεισφορές. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για ορισμένε χώρες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες σε τελική ανάλυση θα πρέπει να εφαρμόσουν την πολιτική αυτή στις περιφέρειές τους. Αλλά γι' αυτό εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν έχουμε επιτύχει ακόμα τον πρέποντα βαθμό της ε, απλοποίησης, δυστυχώς. και θα ήταν απαραίτητο να μπορέσουμε να κάτσουμε και να σκεφτούμε καλύτερα πώς θα μπορέσουμε πράγματι να επιτύχουμε αυτή την απλοποίηση ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν στους σωστούς αποδέκτες το ταχύτερο δυνατό να έχουμε λοιπόν μια τέτοια διαδικασία. Θα μπορούσατε επομένω να μας, ε, να μας εξηγήσετε αν εσεί ω Ισπανική Προεδρία θα κάνετε μία πρόταση για το θέμα αυτό, για αν τουλάχιστον θα διοργανωθούν κάποιε συζητήσει στο Συμβούλιο επί του θέματο αυτού, ότι τουλάχιστον στο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη κοινή βάση σε ό,τι αφορά την προσπάθεια απλοποίηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. And after that you may reply. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο κάποια πρακτικά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Παρουσιάσατε κάποιες ενιολογικές συλλήψεις, οι οποίες μας δείχνουν πώς θα πρέπει να κινηθούμε επέκεινα και του 2013 σε σχέση με αυτές τις βασικές ενιολογικές γραμμές. Θα ήθελα ξέρω αν αυτά είναι μια ισπανική πρόταση ή μια πρόταση της ομάδος εργασίας του Συμβουλίου ή αν αντανακλά αυτά τα οποία προτίθεται να αντιμετωπίσει και να προετοιμάσει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με τη μεταρρύθμιση μετά το 2013. Για μένα είναι σημαντικό να ξέρω αν αυτό είναι θέση του Συμβουλίου ή στοχοθεσία του Συμβουλίου ή γενική συμβαστική θέση ή αν είναι απλώς μια ισπανική θέση. Θα ήθελα επίσης να ξέρω κατά πόσο και πόσο εντατικά θα επιληφθεί η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά, το, του τι θα γίνει μετά το 2013, πόσο συχνά θα συναντείτε αυτή η ομάδα, θα υπάρξουν ενδιάμεσες προτάσεις στο τέλος της Προεδρίας σας, τι ακριβώς προτείνετε σχετικά. Okay, thank you very much. Would you please... Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Το πρώτο ερώτημα που μου έθεσε ο κύριος Φανίστερ Ρόι έχει να κάνει με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό της πολιτικής συνοχής. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι νέοι κανόνες, κάποιες νέες διαδικασίες προκειμένου να θεμελιωθεί αυτή η συνεργασία. Οι συγκεκριμένοι μας στόχοι στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας, που είναι αυτοί οι οποίοι σας συνόψισα και στην αρχική μου παρέμβαση, ε, θα συζητηθούν στην συνεδρίαση που θα γίνει τον ερχόμενο μήνα στη Σαραγώσα και εκεί φυσικά έχει προσκληθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε και τη δική σας τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία Όσον αφορά τώρα στη στρατηγική για το 2020, εμείς ε, θεωρούμε ότι για να δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός μεταξύ πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής για το 2020 είναι να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα και πριν θεωρώ ότι το φόρουμ για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση να προσπαθήσουμε να συζητούμε λίγο περισσότερο πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός είναι η συνεδρία που θα γίνει τον ερχόμενο μήνα στη Σαραγώθα ακριβώς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία όπως ε, σας είπα ε, θα τα συζητήσουμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι προσκεκλημένο και ε, στηριζόμαστε και στην παρουσία σας εκεί. Τώρα, για την απλούστευση. Εδώ θα ήθελα εκ νέου να πω ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε θέση για τη συζήτηση που θα γίνει του Φεβρουάριο και είναι μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας Χωρίς αμφιβολία. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν να θέσουμε, και εδώ σας μιλώ ως διαχειριστής ενός εθνικού προπολογισμού. Στη χώρα μου υπάρχουν τόσο αυστηροί έλεγχοι σαν αυτοί που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και το ίδιο φυσικά θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εμεί είμαστε διαχειριστέ εθνικών προπολογισμών. Και ε, το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχει αυστηρή εφαρμογή σαν αυτή που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο εκτέλεση πολύ ψηλό, Διαχειριζόμαστε προπολογισμού που μπορεί να έχουν κάποιε καθυστερήσει. Ναι, σε κάποιε περιπτώσει υπάρχουν καθυστερήσει, αλλά σε γενικέ γραμμέ είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Και αν το δούμε άλλωστε σε εθνικό επίπεδο, αν τα καταφέρνουμε εκεί, λογικά θα μπορούμε να το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά τα συστήματα εθνικών ελέγχων δεν γεννήθηκαν εκ του μηδενός, ε, προέκυψαν από ένα σύνολο των προσπαθειών και φυσικά το ίδιο κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μαθαίνουμε σιγά σιγά να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Ως εθνικός λοιπόν διαχειριστής ε, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για να βελτιωθούν τα πράγματα χωρίς να αποδυναμηθεί η ισχύ των ελέγχων θα είναι όσο αυστηρή είναι και τώρα, αλλά χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην ε, διακοπεί ο προγραμματισμός. Να μην υπάρχουν χρόνια καθυστερήσεων. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εν μία νυχτή, αλλά φυσικά είναι κάτι το οποίο είμαστε διαδεχμένοι να κάνουμε και θεωρούμε σημαντικό. Και πάλι το Φεβρουάριο στη Σαραγώθα θα εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Τρίτον, ως προς το νόημα της παρέμβασής μου, αυτή είναι η ισπανική πρόταση, αυτήν θα παρουσιάσουμε και στη συζήτηση το Φεβρουάριο στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών. Και αυτή είναι η πρόταση για τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας. Βέβαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν σχετικές εργασίες εν εξελίξη και φυσικά θεωρούμε ότι αυτά θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Η πρόταση όμως που σας παρουσίασα εγώ είναι η πρόταση της Ισπανικής Προεδρίας. Αυτά που σας είπα και στην παρέμβασή μου. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Έχω ακόμα 8 συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Να ζητήσω λοιπόν ότι αν θέλει κάποιος ε, ε, άλλος να προσθεθεί στη λίστα γιατί διαφορετικά ο κατάλογος των αγορτών θα κλείσει. Ο κύριος Μανέσκου. Mulțumesc, uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε uh, Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Αν κατάλαβα καλά, οι στόχοι της Ισπανικής Προεδρίας είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και δείχνουν ότι εστιάζεται στα κυριότερα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο γενικότερα και στην Επιτροπή μας ειδικότερα. Αναφερθήκατε στην κρίση, αναφερθήκατε στις συνέπειες της κρίσης κλπ. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, πέρα από τις προτεραιότητες που παρουσιάσατε εδώ, η Ισπανική Προεδρία για τους επόμενους έξι μήνες αντιμετωπίζει κάποιες άλλες συγκεκριμένε δράσεις έτσι ώστε να στηριχτούν οι χώρες οι οποίες έχουν ε, ιδιαίτερος πληγή από την κρίση όσον αφορά την στρατηγική τώρα του 2020. Δυστυχώς σε αυτήν τη στρατηγική δεν αναφέρονται καθόλου οι τοπικές αρχές. Επιτρέψτε μου λοιπόν κύριε Υπουργέ να σας ρωτήσω Πιστεύετε ότι στους επόμενους έξι μήνες μπορείτε να στρέψετε τη συζήτηση προς το θέμα αυτό, κυρίως ε, μια και η Προεδρία στους στόχους της αναφέρθηκε και στον ρόλο που οφείλουν να παίξουν οι τοπικές αρχές ή οι τοπικοί κυβερνήτες ε, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν μπορεί να επιτύχει η κοινωνία η πολιτική συνοχή. Ο κύριος Ρασάκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Υπουργέ, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα. Αναφερθήκατε εσείς στους ελέγχους. Κατά την άποψή μου, αυτός ε, είναι ένα, αυτά είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία δυσκολεύει ε, περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας ε, για τους μεμονωμένους ελέγχους. Ε, επίσης, όσον αφορά τις στατιστικές μεθόδους, βεβαίως πρέπει να έχουμε όλοι συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Απ' την άλλη πλευρά, δυσκολεύει η κατάσταση για ορισμένους από εμά όταν πρέπει να υποβάλουμε στατιστικά στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τον μηχανισμό για την αύξηση της ελαστικότητας. Κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικές περιπτώσεις βλέπε χρηματοπιστωτική κρίση, πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε αμέσως. Ποια είναι η άποψή σας και ποια είναι τα μέσα αυτά της άμεσης αντίδρασης. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ε, κύριε Αντέλη και μετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, αναλαμβάνετε την Προεδρία στο έτος ε, της καταπολέμησης της φτώχειας. 80 είναι τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι φτωχοί και επομένως κεντρικό ερώτημα αυτό ε, του ε, κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ε, αδικίας που οδηγεί και σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Βεβαίως ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, είναι η, ε, ε, η προβληματική κατάσταση όσον αφορά ε, τους ενεργειακούς πόρους ε, και γνωρίζουμε ότι ε, τα, από το πρόβλημα αυτό απορρέουν μια σειρά άλλων προβλημάτων. Άκουσα προσεκτικά τα όσα μας είπε ο Χωσέ Λουίς Θαπατέρο την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας αγοράς ενέργειας. Όμως το 2007 ο Υπουργός ε, ε, Στέγασης της ε, Ισπανίας είχε εκπονήσει έκθεση σχετικά με την στέγη και την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι πρόσφατα 100.000 ε, φοιτητές διαδήλωσαν με ένα πολύ εύγλωτο σλόγγαν και πάσα νότε νέμος κάσα, δηλαδή τι συμβαίνει, δεν έχουμε σπίτι και επομένως τι έχετε να απαντήσετε σε αυτά. 20 Ensuite, Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσετε για να καταπολεμήσετε συγκεκριμένα και με συγκεκριμένους τρόπους την ένδια και επίσης όσον αφορά ε, την, το ενεργειακό ε, ζήτημα γνωρίζομαι ότι σύντομα θα συναντηθούν στο Τολέδο ε, στις 21 και 22 Ιουνίου δηλαδή του 2010 θα συναντηθούν στο Τολέδο λέγω οι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για την ε, στέγη αλλά και για την ενέργεια και επομένως πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά ε, τα δύο ζητήματα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και επίσης πώς θα αντιμετωπίσετε αυτούς τους τους θύλακες ε, που υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, και είναι θύλακες περιθωριοποίησης ε, και κοινωνικού αποκλεισμού. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Παρισιού αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Και πάλι θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής αν μπορείτε να είσαστε όσο να τον πιο συνοπτικός γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Σοκιάνα. Όπως μου ζητείτε θα είμαι σύντομος. Το πρώτο ερώτημα είναι ποια τα συγκεκριμένα μέτρα ενώπιον της κρίσης θα λάβουμε. Αν είμαστε ρεαλιστές, είναι αδύνατο να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη χρηματοδότηση. Αλλά θα ήταν σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αν μπορέσουμε να εκτελέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα προγράμματα και να εκταμιεύσουμε τους πόρους που έχουμε δεσμεύσει. Να μπορέσουμε όλα αυτά τα ποσά να φτάσουν στον τελικό τους αποδέκτη. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Να μπορέσουμε λοιπόν 100% να επιτύχουμε εκταμίευση στην πολιτική συνοχή. Η περιφερειακή και τοπική συμμετοχή Προέρχομαι από μια χώρα που όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ αποκεντρωμένη και υπάρχει λοιπόν αυτή η όσμωση μεταξύ των θεσμικών οργάνων στα διάφορα επίπεδα που λειτουργεί καλά. Και γι' αυτό συμφωνώ να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια τέτοια θεσμική όσμωση η οποία θα επιτρέψει την τοπική και περιφερειακή συμμετοχή χωρίς τώρα να σας δώσω λεπτομέρειες νομίζω μπορούμε να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν για να υπάρξει η πολυεπιπεδική συμμετοχή. Στατιστική έλεγχη. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικοί για την πολυπικιλία των σχεδίων και μπορεί χωρίς υπερβολικό άχθος να μας βοηθήσουν στην εκτέλεση των ελέγχων. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται τεχνικού χαρακτήρα. Μπορεί να είναι θέμα δειγματοληψίας και στατιστικής τεχνικής, <clears throat> αλλά εμείς έχουμε σαν στόχο να έχουμε την καλύτερη δυνατή δειγματοληψία και να υπάρχει αναλογικότητα στην ε, συλλογή των στοιχείων. Η Ισπανική Προεδρία ελπίζει ότι θα μπορέσει να προωθήσει τα ζητήματα αυτά της περιφερειακής πολιτικής προσαρμόζοντας την ε, πολιτική μας στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ώστε να λειτουργήσουν όλα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στα τελευταία, θέματα, στα τελευταία δύο θέματα που αναφέρατε επιτρέψτε μου να μην παρέμβω γιατί δεν είναι δικά μου θέματα. Το θέμα της επισφαλούς παροχής ενέργειας και της επισφαλούς στέγασης. Κατανοώ ότι αυτά είναι σημαντικά θέματα, αλλά υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι της Ισπανικής Προεδρίας που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά προς την κατεύθυνση ακριβώς που αναφέρατε. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργό τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που θα πρέπει να αποδώσουμε στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά ανασφάλειας στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Αλφονσί μετά Λάρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ή τρία ερωτήματα να θέσω. Πρώτα απ' όλα, η Ισπανική Προεδρία πώς προτίθεται να δράσει στο επίπεδο της πολιτικής συνοχής ώστε οι χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό όχι μόνο να μειωθούν λόγω της κρίσης του προπολογισμού, αλλά να ενισχυθούν και στο μέλλον. Γιατί αυτό είναι το βασικό για να επιτύχουμε την, την ανάπτυξη μιας πολιτικής, χρειαζόμαστε οικονομικά μέτρα. Και τώρα υπάρχει όλη η προβληματική στις λεγόμενες μακροπεριοχές. Υπάρχει η μακροπεριοχή της Βαλτικής με επί, επί της Σουηδικής Προεδρίας που προωθήθηκε η περιοχή του Δούναβη που θα προωθηθεί από την Ουγγρική Προεδρία εγώ ως προχώμος από την Κορσική θα ήθελα η Ισπανική Προεδρία να αναπτύξει μια μακροπεριοχή, μια μέγα περιοχή που να καλύπτει τη Μεσόγειο. Γιατί σήμερα που μιλάμε <clears throat> ακόμα δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει εμπορέματα μεταξύ Κορσικής και Μασαλίας. Έρχονται τα καμιόνια στη Μασαλία, πηγαίνω στη Γένοβα, ένας από τους πιο ε, και κορεσμένους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης για να μπορέσουν να πάνε στην Σαρδινία. Πώς λοιπόν σκεφτόσαστε να, να ε, εισαγάγετε και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Σας δίνω μια γελιογραφική, αν θέλετε, κατάσταση αυτό που είπα προηγουμένως για τη Σαρδινία και την Κωσική. Επίσης, θα θέλαμε να υπάρξει μια συζήτηση σε σχέση με τα κριτήρια που εφαρμόζεται για το ΑΕΠ κατά κεφαλήν. Μήπως μπορούμε να ξεπεράσουμε το κριτήριο μοναχα του ΑΕΠ ως γνώμονα της περιφερειακής πολιτικής και να δούμε και ευρύτερους δείκτες. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση. Την άποψή σας για την έκδοση Μπάρκας. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι δεν θα έχουμε περισσότερα χρήματα, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε πιο αποδυτικά. Στην έκθεση του καθηγητή Μπάρκας υπάρχει ένα πυλώνα υπαριθμών 10, στον οποίο προτείνεται σε κάθε κράτο μέλος να δίνει μία δήλωση ε, κάθε τρία χρόνια για την αποτελεσματικότητα τη χρήση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αφετέρου, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το 2009 μελέτες για τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων σε παραμέτρους όπως είναι η ανεργία, το ισοζύγιο πληρωμών, η αύξηση του ΑΕΠ, εισαγωγές και εξαγωγές. Η ερώτησή μου είναι εξή. Στην Επιτροπή Προπολογισμών πιέζουμε να γίνει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προπολογισμού, ώστε να είναι σαφές πώ χρησιμοποιούν τα κονδύλια γενικώ και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Τι έχει να προτείνει η Ισπανία για αυτό το σκεπτικό ε, της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων, των περιφερειακών ταμείων και των προτάσεων του καθηγητή Μπάρκα. Thank you very much. Mr. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός κύριος Οκάνια ε, μας είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι όσον αφορά την ε, πολιτική συνοχή ε, η Ισπανία άλλαξε πρόσωπο όπως το είπε και ο κύριος Ταπατέρο βάση της ε, ε, πολιτικής ε, συνοχής και βάση της σωστής χρηματοδότησης που είχαν τότε όμως γνωρίζομαι ότι στις νέες χώρες η οικονομική πολιτική θα είναι τελείως διαφορετική 2005 και 2007 ε, τα ε, πράγματα όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με τα ταμεία συνοχής διαπραγματεύτηκαν και συζητήθηκαν ε, και βρέθηκαν κάποιοι τρόποι και κάποιες παράμετροι. Όμως ρωτώ Πώς πιστεύετε ότι θα λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά το μέλλον ε, των, ε, ε, της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική αυτή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι θα αποτελέσει τμήμα της νέας δημοσιονομικής πολιτικής και βεβαίως το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και φυσικά μας ενδιαφέρει με ποιο μηχανισμό θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Thank you Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Το πρώτο ερώτημα ήταν οι ε, ήδη υπάρχονται σε δεσμεύσει στον προπολογισμό και πώς σκοπεύουμε να τις στηρίσουμε. Και εδώ να πω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Οι δημοσιονομικές προοπτικές ε, είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των προβλημάτων των διαφόρων περιφερειών και των διαφέρων χωρών ε, που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, ε, αυτό να διαμφισβήτη το. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και αυτό είναι προτεραιότητά μας, οι δεσμεύσεις αυτές να εκτελεστούν με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε επίση τη διαμεθοριακή συνεργασία, διότι αυτό είναι αυτό το οποίο συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά την άποψή μας αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σεβόμενοι την ε, ε, χρηματοοικονομική ιδιαιτερότητα. Οι πόροι είναι λίγοι και οι μακροπεριοχές δεν ε, σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια που θα έχουμε, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να ξοδεύουμε καλύτερα και να γίνεται καλύτερη κατανομή των πόρων που διαθέτουμε. Προτείνεται την αλλαγή δικτών. Να έχουμε άλλους δείκτες και όχι μόνο το ΑΕΠ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Γιατί όχι, να μην δούμε και άλλα μέτρα. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζουμε και τι περιορισμούς έχουμε στην εισαγωγή ε, κριτηριών τα οποία θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικά και δι, διότι η θα είναι ε, πολύ πιο εύκολο να τα επικρίνει κάποιο και μπορεί και να μην είναι αντιπροσωπευτικά, να μην αντικατοπτρίζουν το σύνολο, αλλά να είναι πιο ομογενεί ε, σε κάποιε άλλε χώρε. Μπορεί να είναι δηλαδή πιο εύκολο να κάνουμε σύγκριση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Να είμαστε πιο ακριβείς αλλά πιο υποκειμενικοί και να έχουμε συνένεση ή να έχουμε κάποια πιο απρά, απλά στοιχεία τα οποία ναι μεν χάνουν κάποιες πληροφορίες αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να τα παρακολουθήσουμε και να τα συγκρίνουμε. Κάθε θέμα έχει διαφορετικές συνιστώσεις και θα πρέπει να δούμε διαφορετικές μεταβλητές. Ε, Παραδείγματο χάρη, αν σκεφτώ τις ισπανικές περιφέρειες, ε, σε κάποιες έχουμε ε, μικρή πυκνότητα πληθυσμού, σε κάποιες έχουμε μεταναστευτικές ροές που δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και στην παιδεία και δημιουργούν και επιπλέον ε, κόστος ε, στην υγεία και στην παιδεία. Σε άλλη περιφέρεια έχουμε το θέμα της απομόνωσης γιατί είναι νησιά και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και καταλαβαίνετε ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να τη σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο διότι κάθε μία έχει διαφορετικές δομές κόστους. Φυσικά είναι πολύ χρήσιμο να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε δείκτες που θα είναι πιο ελαστικοί και θα αντικατρίζουν τα πάντα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και μήπως ε, περιπλέκοντας τόσο πολύ τους δείκτες θα έχουμε μια πολύ πιο υποκειμενική και πολύ πιο δύσκολη συζήτηση και δεν θα μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα. Ναι, μεν λοιπόν συμφωνώ στο να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της ε, πολιτικής συνοχής, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε λίγο λογικοί και να ξέρουμε ότι η απόλυτη ακρίβεια μπορεί και να μην είναι πανάκια. Διότι πρέπει να έχουμε δείκτες που θα είναι συγκρίσιμοι και που θα είναι γενικώς αποδεκτοί. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο και θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Οι επιπτώσει τη πολιτική συνοχή ε, τελικά φαίνονται στον προπολογισμό, στον εθνικό προπολογισμό. Αν μια χώρα δεν έχει ανάπτυξη είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να υποστηρίξει και την περιφερειοποίηση. Τίποτα άλλο ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ μικρή, σύντομη ερώτηση, κύριε Μαδόρο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο μάλλον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτάκι και θα ήθελα να αναφερθώ μονάχα σε δύο θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στον καθορισμό κάποιων μεταβατικών περιόδων στις οποίες ε, οι περιφέρειες ενδεχομένως ε, θα έχουν κάποια απόσταση από τους στόχους συνοχής. Αναφερθήκατε ε, σε τέτοιες μεταβατικές περιόδους έτσι ώστε να φτάσουμε σε κατάργηση της χρηματοδότησης. Σε ποιοι θα είναι όμως οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι θα αποτρέψουν τον κίνδυνο ανοίγμα ανοίγματο της ψαλίδας και επομένως διεύρυνση των αποκλήσεων μεταξύ των περιφερειών. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που είπε και η κυρία Μανέσκου, δεν υπάρχει καλό συντονισμός ανάμεσα στο Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Εσείς ε, αναφερθήκατε στις ε, καλές σχέσεις ε, που πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις χώρες ανάμεσα στις περιφέρειες και βεβαίως το παράδειγμα της Ισπανίας είναι πολύ καλό γιατί εσείς έχετε μια αποκεντρωμένη χώρα με καλές σχέσεις. Όμως πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των περιφερειακών ταμείων Ταμείων έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερη συνεργασία. Thank you very much, ε, ε. Ευχαριστώ, κύριε Κωστές. Τελευταίο ερώτημα. Κύριος Κορτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Οκάνια, θέλω να χαιρετήσω την παρουσία σας, την σαφή σας παρουσίαση και τις σαφείς εξηγήσει που δώσατε για το έργο της Ισπανικής Προεδρίας. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας θέσω δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα και σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, που έχετε αναφέρει ήδη τα θέματα αυτά, μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η αντιμετώπιση των λεγόμενων μεταβατικών περιοχών και δεύτερον, ποια ήταν η συμβολή τη πολιτική συνοχή του επίτευξη των στόχων τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ πολύ και ο γύρος Ορό για το τελευταίο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, είδα στο πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας να υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία αφορούν τις υπερπεριφερειακές περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές. Θέλω να θέσω λοιπόν μερικά ερωτήματα για το θέμα αυτό. Με ποιο τρόπο η Ισπανική Προεδρία <clears throat> θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών. Επίσης, αν θέλει η Προεδρία να εφαρμοστεί της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπερπεριφερειακές περιοχές ένα ατού για την Ευρώπη, όπως αναφέρει ο τίτλος της. Πώς θα προχωρήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει το στόχο αυτό και ποια μέτρα προβλέπετε εσείς να εφαρμόσετε και τέλος ένα ακόμα ερώτημα για τις υπερπεριφερειακές περιοχές θεωρεί η Προεδρία ότι θα πρέπει να εργαστεί για μια καλύτερη ενσωμάτωση των περιοχών αυτών στην θαλάσσια λεκάνη στην οποία βρίσκονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Thank you very much. Minister, you have the floor. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Δύο λεπτά έχω να χάσω για να απαντήσω σε έξι ερωτήσεις. για τις μεταβατικές περιόδους για τις μεταβατικές περιοχές μάλλον. Η ιδέα ήταν να μην υπάρχουν απότομες αλλαγές σε ό,τι αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ό,τι αμφισβητεί η εμπειρία μας με το phasing in και phasing out των περιοχών στην τωρινή περίοδο προγραμματισμού είναι ότι έγινε ο προγραμματισμός με τέτοιο τρόπο ώστε ήταν δύσκολο να υπάρξει σωστή εφαρμογή των ε, πόρων στο μέλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι θα επανέλθει το θέμα αυτό στην μελλοντική περίοδο προγραμματισμού, είναι απαραίτητο λοιπόν σε αυτές τις περιοχές που είναι σε μεταβατική θέση να υπάρχει μια πιο ομαλή κατανομή πόρων μέσα στον χρόνο. Επίσης, για να αποφύγουμε συνέχειες, όπου για λόγω μικρής αύξησης του κατακεφαλήν ΑΕΠ μια περιοχή αλλάζει στόχο, είναι απαραίτητο να έχουμε μια πολιτική βαθμία ώστε να έχουμε και την σωστή προσοχή στην διαδικασία ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Για το θέμα της διακυβέρνησης τώρα, για το ποιος θα πρέπει να συντονίζει την κατανομή των πόρων όταν υπάρχουν εξουσίες σε διάφορα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό στην πράξη είναι ότι στην πράξη αυτό που έχει λειτουργήσει καλύτερα είναι η κατανομή σε επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο εθνικού κράτους. Δεν μπορεί λοιπόν καμία κατανομή να παραγνωρίζει την ύπαρξη κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Sobre, sobre las, ε, σε σχέση με τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Τον Μάιο θα γίνει μια ειδική συνδιάσκεψη για τα θέματα αυτά και εκεί θα θέλαμε να προωθήσουμε τη συζήτηση για τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Είναι πολλές χώρες της Ευρώπης που έχουν τέτοιες υπερπεριφερειακές περιοχές, αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα οι εφαρμογές των κοινοτικών ταμείων στις περιοχές αυτές. Και τα προβλήματα αυτά είναι περισσότερο προβλήματα πρακτικά και όχι οργάνωσης και σχεδιασμού, αλλά το Μάιο θα γίνει πράγματι αυτή η ειδική συνδιάσκεψη για την περίπτωση των υπερπεριφερειακών περιοχών. Κύριε Κορτές, αναφερθήκατε κι εσείς στις περιοχές, στις που βρίσκονται σε μία μεταβατική φάση Και πάλι σας λέω ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστά. Έχουμε δεχτεί τη βασική αρχή να μην υπάρχουν έντονες ασυνέχειες λόγω μιας μικρής αλλαγής από μια δημοσιονομική περίοδο προοπτικών μέχρι την επόμενη. <clears throat> να υπάρξει λοιπόν μια δυνατότητα απάλυνσης αυτών των ασυνεχειών. και ο στόχος της πολιτικής συνοχής προφανώς είναι να εξασφαλίσει την σύγκληση μεταξύ περιοχών και περιφερειών και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Νομίζω ότι έχουμε το σωστό σύστημα και χρειάζεται βέβαια να προβούμε σε ένα fine tuning, δηλαδή σε μια διαρρύθμιση για τις μεταβατικές περιόδους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι εξυπηρετεί το στόχος της σύγκλησης και της ανταγωνιστικότητας. Και πάλι σας λέω δεν πρέπει να αλλάξουμε τις κύριες γραμμές, τις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά να κάνουμε λεπτομεριακές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ, την παρουσίασή σας, τα σχόλια και τις ε, ε, απαντήσεις που δώσατε και βεβαίως ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, για τη συζήτηση που κάναμε. dear colleagues, shall we continue? Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. Okay. Yeah. Miguel, yes? you want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα ένα δοκιμαστικό ε, της ε, ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Ε, ψήφισαν όλοι. Για μία ακόμα φορά. Ας ασκηθούμε λίγο. Ψήφισαν όλοι. Όχι ακόμη. It Δυστυχώς δεν έχω την κάρτα μου, κύριε Πρόεδρε, μαζί μου. Εντάξει, κύριε Κέλλη, θα σας ε, μετρήσουμε, θα σας προσμετρήσουμε την ψήφο σας, τέλος πάντων. Να πούμε τώρα ότι ψηφίσαμε όλοι πέρα τη ψηφοφορία πάρα πολύ ωραία.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 Προχωράμε λοιπόν στο σημείο 5, έκθεση σχετικά με την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής ε, όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης. Εισηγητής ο κ. Σαλβατόρε Γκαρόνα. Έχετε λοιπόν μπροστά σα ε, τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να ε, ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω χάσει, δεν την έφερα μαζί μου την κάρτα μου, δεν έχω φέρει την κάρτα μου μαζί μου, γι' αυτό λοιπόν, ε, εν πάση περιπτώσει, έχω καταψηφίσει. Okay. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το αποτέλεσμα. Ε, νόμιζα ότι όταν ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ θα πρέπει να μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα στι οθόνε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ναι, έχετε δίκιο. We go to the amendment number two. Περνάμε λοιπόν στη τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Βαν λέει. Κύριε Πρόεδρε, ίσως πρέπει να θέσω την ερώτησή μου ευθέως. Θέλω να δω το αποτέλεσμα της προηγούμενης ηλεκτρονικής πληροφορίας. Τα στοιχεία μπορείτε να μας τα πείτε. Κατάλαβα ότι απορρίφθηκε η τροπολογία, αλλά θέλω να ξέρω τους αριθμούς. Okay, 22. 22 ψήφοι κατά, 17 υπέρ. Συγγνώμη για την παράληψη. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία ή μάλλον όχι, να ψηφίσουμε έτσι. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. In favor. Το επόμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 5, 6, 3, 4 καταπίπτουν. Προχωράμε τώρα. Τροπολογία υπαριθμών 7. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της, του τροπολογίας 7. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Και εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τμήμα 3 να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Προφορική τροπολογία του ΕΛΚ ε, η οποία θέλει να αντικαταστήσει το develop το, το reinforce υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τμήμα 2. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 3. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι σαφές. Τροπολογία 16. Πρόκειται εδώ, για προφορική τροπολογία του κυρίου Καντέκ που θέλει πριν από τις αρχές να ε, βάλουμε το επίθετο τοπικές υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 προφορική τροπολογία του εισηγητού που θέλει να διαγράψει τη λέξη instrument, εργαλείο, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19, 19, 21 και 22 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε επομένως στην τροπολογία 23. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Προφορική τροπολογία από τους πράσινους. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ. Μάλλον όχι, λέει ο Πρόεδρος. Ψήφισαν όλοι Πέρα της ψηφοφορίες. Δεκαέξι ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Επομένως απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, 17 κατά και επομένως εγκρίνεται. Άρα, κυροπολογίες 27, 29, 30 και, 20, και 30 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 28. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν επί της 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 31 ψήφι υπέρ, 8 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 34. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 37 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η τροπολογία 35. Προχωράμε λοιπόν στην τροπολογία 38. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επομένως, καταπίπτουν η τροπολογία 39 και 42 και ψηφίζουμε την τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές. Δεν είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Επομένως, ε, ενεκρίθη η τροπολογία. Ψηφίζουμε επί της νομοδοτήσεως. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Επομένως ε, έχουμε 29 ψήφους υπέρ 8 κατά, άρα ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο καρόνα. Συγγνώμη, πρέπει να απουσιάσω για μισή ώρα. Θα συνεχίσει ο συνάδελφος, ε, ο κύριος Πέπερ, για τις επόμενες ψηφοφορίες. Ja, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με την ψηφοφορία για την έκθεση των <clears throat> χρηματοοικονομικών συμφερόντων αγώνας κατά της ε, απάτης. Ετήσια έκθεση 2008. Ψηφίζουμε <clears throat> την παραγραφό 1. Τροπολογία 1. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκπίπτουν κατά συνέπεια οι τροπολογίες 2, 3 και 4. Ψηφίζουμε τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 13 ψήφοι κατά, γίνεται δεκτή. Τροπολογία 6. Έχει αποσυρθεί όμως. Ψηφίζουμε την 7. <clears throat> Ψήφοι υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, η 7 έχει εκπέσει, διότι έχει εγκριθεί η 5. Σωστά. Μεγάλο το δίκιο σας. Τροπολογία 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 <clears throat> ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ελέγχου για την 13. Άρχεται. Πέρας. 23 υπέρ, 17 κατά. Γίνεται δεκτή επομένως. 14 <clears throat> ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ψήφι υπέρ ηλεκτρονικά μάλλον. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρα ψηφοφορία. 38 υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Ματσόνη. Το επόμενο σημείο πρέπει να ξεκουραστούν τα μηχανήματα λιγάκι, λέει ο πρόεδρος. Είναι σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με εισηγητρία την κυρία Κρέελ. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5. Πέρας ψηφοφορίας. Είκοσι, είκοσι, απορρίπτεται, επομένως λόγω ισοψηφίας. Α, δεν είχατε κάρτα όμως. Ο κύριος Κέλλη ήταν υπέρ, οπότε εγκρίνεται. εγκρίνεται ίσα ίσα στην τρίχα. Τροπολογία 6, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 7, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική μορφή, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μία ισχυρή πλειοψηφία. 38 ψηφί υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Κρέελ. Προχωρούμε λοιπόν. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι θα συνεχίσουμε και αύριο στις 9. Το λέω γιατί ορισμένοι δεν είχαν τα ακουστικά τους. Και αυτό είναι αντίθετα από τις ενδείξεις που είχαμε στην αρχή στην ατζέντα μας, αλλά αύριο πράγματι συνεχίζουμε την ημερησία διαταξή μας. Το τονίζω. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 8. Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, έλεγχος υγείας της γεωργικής πολιτικής. Η συγκήτρια μας είναι η κυρία Φεραγκούτ και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης της. Παρακαλώ κυρία Φεραγκούτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάζουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης στην ίδια άγουσα που είχε ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτουσίας Επιτροπή, Επιτροπή Γεωργίας, γνωρίζοντας ότι αυτές οι περιοχές θεωρούνται περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και καλύπτουν το 80% της ε, γεωργικής επιφάνειας. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένα μειονεκτήματα και ορεινές περιοχές, αλλά εμείς θα εστιάσουμε στις ενδιάμεσες περιοχές οι οποίες έχουν φυσικά μειονεκτήματα και αυξημένο ε, ποσοστό ε, απομάκρυνση του πληθυσμού από τις υπόλοιπες περιοχές. Ε, τα θέματα που θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες θα είναι πολύ σημαντικά ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχουν για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα η γνωμοδότηση βασίζεται στο εξή. Πρώτον είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον μελλοντικό καθορισμό των αποζημιώσεων να μειωθούν ουσιαστικά οι ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις βοήθειες που δίνονται ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουμε να τηρήσουμε το βασικό στόχο που είναι η αρχή της συνοχής. περνάμε από τα 16 ευρώ αναστρέμα που έχουμε στην Ισπανία στα 212 ευρώ αναστρέμα που έχουμε στο Βέλγιο. Ε, σε κάθε ε, χώρα έχουμε μεγάλες διαφορές, γι' αυτό και ακριβώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, υπερτώνησε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε σήμερα είναι το θέμα της φυγής του πληθυσμού. Της μείωσης του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή ε, προτείνει να μην λαμβάνεται υπόψη αυτό το κριτήριο της μείωσης του πληθυσμού και αυτό που θέλουμε εμείς είναι το κριτήριο αυτό να λαμβάνεται υπόψη ε, ως ε, τελική ρύθμιση, διόρθωση, διότι ε, η μείωση του πληθυσμού σαφώς επιδεινώνει τα μειονεκτήματα που έχουμε και φυσικά υπάρχει και μεγάλη αποκέντρωση, ε, μάλλον συγγνώμη, συγκέντρωση πληθυσμού σε άλλες ε, σε αστικές περιοχές. Υπάρχουν ε, αυτοί που θέλουν ε, να κάνουν ε, μια ριζική μεταρρύθμιση των ενδιάμεσων αυτών περιοχών και άλλοι που θέλουν να κρατήσουν κάποια, κάποιο μέτρο. Και αυτή λοιπόν η διόρθωση που θα γίνει για τη μείωση του πληθυσμού θα είναι πολύ σημαντική. Επίση, θέλουμε να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίοδο που θα δίνεται για να γίνει προσαρμογή για αυτή τη νέα ταξινόμηση, τη νέα κατηγορία των ενδιάμεσων περιοχών και να τους δοθεί μια μεταβατική περίοδος ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε και κάποια μέτρα ε, τα οποία θα μετριάσουν την κατάσταση. Ε, κάτι ακόμα που ζητάμε είναι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να ρωτούνται, όπως επίσης και οι ενδιαφερόμενοι αγροτικοί σύλλογοι. Ε, έχουν δοθεί οκτώ κριτήρια επιστημονικού χαρακτήρα. Αυτά τα κριτήρια τα έδωσε η Επιστημονική Επιτροπή και είναι βιοφυσικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος χάρτης για να καθορίσει ποιε θα είναι οι περιοχές που θα προκύψουν και καλό θα ήταν να ακούσουμε και την άποψη των διαφόρων αρχών σε αυτή τη διαδικασία, ε, τόσο των τοπικών όσο και των περιφερειακών αρχών. Ένα ακόμα στόχο ο οποίο ετέθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο ήταν η ανισότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε πότε μια περιοχή θεωρείται μια ενδιάμεση ή όχι περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 κριτήρια ε, λόγω των μεγάλων ε, περιθωρίων διακριτική ευχέρειας που έχουν τα κράτη-μέλη και αυτό είναι αυτό το οποίο κατήγγειλε κατά βάση το ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να πλουστεύσουμε το καθεστώς και να καθορίσουμε ε, ε, αντικειμενικά κοινοτικά κριτήρια. Αυτή είναι η θετική πτυχή της πρότασης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει εδώ να επενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν και κάποιο περιθέωριο ευελιξίας, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν και κάποια εθνικά κριτήρια ε, με στόχο να προσαρμόσουν το σύστημα στην ε, ε, υπάρχουσα κατάσταση. Για να επανέλθω τώρα και σε αυτούς τους λεπτούς χειρισμούς τους οποίους αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμαστε και στις περιοχές ε, στις οποίες οποίες οι τεχνικές πρόοδοι έχουν καταφέρει να υπερβούν κάποια φυσικά μειονεκτήματα και φυσικά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος αυτών των μεγάλων τεχνικών ε, αλλαγών και τις περιοχές τις οποίες ε, οι εναλλακτικές περιοχές, καλλιέργειες είναι περιορισμένες, για παράδειγμα, ή η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών μέσων. Εγώ να σας πω επίσης ότι ως συντάκτηρα της γνωμοδότησης ε, σας περιέγραψα λίγο τηλεγραφικά ποιες είναι οι προτάσεις του σχεδίου γνωμοδότησης, αλλά υπάρχουν και μία σειρά από τροπολογίες και να πω ότι θα κάνω και εγώ τροπολογίες στην ίδια μου τη γνωμοδότηση, διότι πραγματικά θεωρώ ότι πρόκειται μια ευκαιρία, για μια ευκαιρία να ε, τονίσουμε όλες αυτές τις περιοχές ε, με συγκεκριμένα φυσικά μειονεκτήματα, να λάβουμε υπόψη δηλαδή την πραγματικότητα, την υπάρχουσα κατάσταση, τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, η οποία είναι λίγο αμφίσιμη, δεν περιλαμβάνει ε, τις περιοχές το, νησιωτικές, ούτε τις υπερπεριφερειακές περιοχές ε, και είναι τόσο συγκεχημένος ο ορισμός για τις περιοχές με φυσικά νονεκτήματα που δεν περιλαμβάνει πλέον τις ε, νήσους. Επομένως προτείνεται και μια τροπολογία για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε το σημείο αυτό. Ε, το γεγονός ότι αποκλείστηκαν αυτές οι περιοχές ε, είναι Σημαίνει ότι η Μενόρκα στις Βαλεαρίδες Ρήθου αποκλείστηκε από βοήθειε, τι οποίες λάμβανε ιστορικά, για ιστορικούς λόγους. Ε, θα κάνω λοιπόν κάποιες τροπολογίες για να βελτιώσω το κείμενο της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Φεραγκούτ. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου. 22 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση και θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Αλφόντς είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενη για αυτή την έκθεση. Κριτήρια όπως η νησιωτική κατάσταση αλλά και επίσης η μικρή πυκνότητα πληθυσμού και η απόσταση από τα κέντρα παραγωγής είναι πράγματι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί είναι σημαντικά μειονεκτήματα. Εξάλλου, θα δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα να υπάρξουν τοπικές προσαρμογέ, να υπάρξει μια ευκαμψία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών και τέλος θα ζητήσουμε να υπάρξει αναβάθμιση των αρρωγών προς τις πιο μειονεκτικέ περιοχέ. και επίση να τονίσουμε ότι πρέπει να είναι <clears throat> οι ίδιοι οι παραγωγοί οι οποίοι θα πάρουν τις βοήθειες αυτές, γιατί σε πολλές περιοχές υπάρχει μια κερδοσκοπική δραστηριότητα που γίνεται σε βάρος των παραγωγών, σκέφτομαι για περιοχές όπως η Σκοτία χάρη, γίνεται σε βάρος αυτών οι οποίοι ασκούν πράγματι την παραγωγική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ίδια την παραγωγική διαδικασία και όχι απλώς αυτούς οι οποίοι επενδύουν χρήματα στις διαδικασίες αυτές. Ακολουθεί ο κύριος Ογώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή έχει σαν στόχο να προσαρμόσει τα νέα κριτήρια που θα αφορούν στις περιοχές οι οποίες έχουν φυσικά μειονεκτήματα. Έχουμε καθορίσει οκτώ κριτήρια τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι η συγγήτρια έχει δώσει ήδη μια θετική απάντηση στο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω, θα ήθελα να έχω και την επιβεβαίωση από αυτήν. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεθνής Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένας χάρτης των περιοχών που θεωρούνται ότι έχουν φυσικό μειονέκτημα. <clears throat> Χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, αλλά επίσης και τα υπερπεριφερειακά διαμερίσματα της ε, Γαλλίας που θεωρούνται στο σύνολό τους ως επιλέξιμα για το ταμείο αυτό. Το ερώτημά μου είναι αν η έγκριση αυτών των νέων κριτηρίων θα τροποποιήσει την κατάσταση που αφορά τα διαμέρισματα αυτά. Τελευταία παρατήρηση. Μεταξύ των κριτηρίων αυτών, μήπως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ως ε, γνώμονα καθορισμού περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα τις περιοχές που τα εδάφη τους είναι ιδιαίτερα ρυπασμένα από χημικούς παράγοντες ή ουσίες που είναι βλαβερές από, από, για την ανθρώπινη υγεία. Ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και αυτό το κριτήριο λοιπόν. Επίσης ερώτημα από τον κύριο Ομπεαμάια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κυρία εισηγήτρια αναφέρθηκε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά την ποιοτική αναβάθμιση των περιφερειών και αυτό θα γίνει μέσω του καλύτερου τεχνικού εξοπλισμού τους, των υποδομών τους. Αλλά η το θέμα της ε, υποδομής και των τεχνικών εξοπλισμών μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την αφή, την αηφορία. Να σας δώσω σαν παράδειγμα τη χρήση βαρέων φορτηγών, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μια τεχνική βελτίωση, αλλά παράλληλα οδηγούν και σε πίεση προς το περιβάλλον και επομένως με τον τρόπο αυτό οδηγούν σε μια δυσκολία σε επίπεδο οικολογικό. Επίσης το θέμα της υδροδότησης. Αυτό φαίνεται καταρχήν ότι είναι θετικό, να υπάρχει καλύτερη χρήση λοιπόν των υδάτων, αλλά όλα αυτά οδηγούν σε απερίμωση των περιοχών και επομένως ούτε και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια ευφυής τεχνική οδός. Επομένως δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτόματο ότι η δημιουργία τεχνικών υποδομών είναι ο καλύτερος δρόμος για να εξασφαλίσει την αηφορία της οικονομικής δραστηριότητας σε μια περιοχή. Έχουμε άλλους δύο μιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το πολύ καλό αυτό σχέδιο γνωμοδότησης. Μπορώ να συμφωνήσω με τα έξι σημεία τα οποία αναφέρατε. Σημαντικά σημεία είναι αυτά για να βελτιώσουμε την περιφερειοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδιος για τα σημεία 2 και 3 θα ήθελα εδώ να σταθώ και να θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο λέτε στο σημείο 2, όπου μιλάτε για, την, για τον αποπληθυσμό ορισμένων περιοχών και θέλετε αυτό να αποτελέσει κριτήριο πόσο συγκεκριμένο ή πόσο σχετικό είναι το στοιχείο αυτό της μείωσης του πληθυσμού μεταξύ των άλλων κριτηρίων. Έχετε την ίδια άποψη όπως και η Κομισιόν για το θέμα αυτό και για το σημείο 3 θέλω και εδώ μία διευκρίνηση. Μιλάτε για μια μεταβατική περίοδο, αλλά πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβατική περίοδος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολένιτσακ το τελευταίο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σημειώσω ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται θα υποστηρίζει αυτές τις ενδιάμεσες μειονεκτικές ζώνες ε, στοχεύει απευθείας ε, στο Γεωργό. Μιλάμε για υποστήριξη αναστρέμα για μικρές εκτάσεις ε, τις τάξεις των 100 ή 150 ευρώ, τουλάχιστον για τα νέα κράτη-μέλη είναι τόση βοήθεια. Και να επισημάνω επίσης ότι κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας στην παραγωγή. Δεν συνεισφέρει σε καμία περίπτωση για να διατηρηθεί ο πληθυσμός μιας περιοχής και για να αποτρέψει την ε, ε, μείωση του πληθυσμού. Στο μέλλον λοιπόν ε, κάποια νέα προγράμματα για, την, για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μέτρα και για τις τοπικές αρχές αλλά και για τους γεωργούς οι οποίοι από κοινού θα ετοιμάσουν κοινούς στόχους. Ίσως ε, αξίζει τον κόπο να ε, το επισημάνουμε αυτό για το μέλλον, ώστε τα κονδύλια από το πρόγραμμα αυτό να μην διοχετεύονται απευθείας ε, στους γεωργούς, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε τουλάχιστον για την Πολωνία ε, καταμερισμό των κονδυλίων σε πάρα πολύ μικρέ εκμεταλλεύσεις και επομένω δεν μπορεί να γίνει τίποτα από πλευρά υλοποίηση των στόχων αυτού του προγράμματο. Παρακαλώ λοιπόν σημειώστε το αυτό. Θα... Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σα ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Έχει ζητήσει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ότι υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο ότι είναι έτοιμο να λάβει το λόγο και θα δώσω μετά το λόγο στην κυρία Φεραγκούτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια δήλωση για τα θέματα αυτά. τα μέτρα αυτά για τις μειορεκτικές περιοχές πρέπει να ατενιστούν στο πλαίσιο της γενικής χωροταξικής και περιφερειακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα των περιοχών που έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους όπως ε, αναφέρθηκε προηγουμένως και αναφέρθηκε η δυνατότητα <clears throat> να υπάρξει και μια στρατηγική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Η πολιτική αυτή ασκείται φυσικά από τα περιφερειακά προγράμματα και μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η υποστήριξη των φυσικά μειονεκτικών περιοχών είναι ένα από διάφορα μέτρα. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η προβληματική σε σχέση με την υποστήριξη των περιοχών αυτών. Ο στόχος αυτής της υποστήριξης είναι σαφής και η νομική βάση είναι σαφής ότι αφορά τις φυσικά μειονεκτικές περιοχές και όχι άλλες περιοχές που μειονεκτούν για άλλους λόγους, όπως οι περιοχές που έχουν απογυμνωθεί από τον πληθυσμό τους. Και επειδή υπάρχει μια πολυπληθώρα και πολυπικιλία εθνικών κριτηρίων σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, εμείς έχουμε προσπαθήσει να καταλήξουμε σε κοινά κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά από μια μακρά διαδικασία ε, διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη, με τους επιστήμονες του τομέα, και με το ευρύ κοινό, σε μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε κριτήρια τα οποία τώρα θα πρέπει να τύχουν δοκιμασία στα κράτη-μέλη. <clears throat> το ερώτημα τώρα, σε ποιο βαθμό πρέπει να συνεχίσουν περιοχές οι οποίες μέσα από διάφορα μέτρα έχουν ξεπεραστεί, περιοχές δηλαδή οι οποίες στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες αλλά σήμερα με την αποστράγγιση παραδείγματος χάρη ε, ελοδών περιοχών μπορούν να είναι παραγωγικές περιοχές <clears throat> αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι σωστό να υπάρχει υποστήριξη μειονεκτικών περιοχών, αλλά πρέπει να θέσουμε το ερώτημα γιατί περιοχές όπου υπάρχει επαρκές εισόδημα για τους παραγωγούς και όπου υπάρχει οικονομική δραστηριότητα επαρκής, γιατί πρέπει να θεωρούνται και αυτές ότι καταλέγονται στις περιοχές ε, που είναι φυσιο, φυσικά μειονεκτικές. Όλη αυτή η προβληματική λοιπόν πρέπει να εξεταστεί ώστε να μπορέσουμε <clears throat> να δικαιολογήσουμε την λήψη μέτρων υπέρ αυτών των περιοχών. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την ε, χρήση εθνικών κριτηρίων για την οριοθέτηση αυτών των περιοχών. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια σημεία επίκρισης από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Αν παραδείγματος χάρη εφαρμοστούν κριτήρια του ΦΕΝΤΕΡ για την ε, οριοθέτηση των περιοχών αυτών, Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα να εφαρμόσουμε τη λογική των φυσικά μειονεκτικών περιοχών, αλλά η χρήση εθνικών κριτηρίων οριοθέτησης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταβατικές περιόδους. Εμείς είμαστε ακόμα στη μέση της διαδικασίας αυτής και τα κράτη-μέλη θα πρέπει προηγουμένως να μας δώσουν τα αποτελέσματα τα οποία, στα οποία θα καταλήξουν με μια προσωμείωση των κριτηρίων και των αποτελεσμάτων τους και μετά θα πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω διαβούλευση με τα κράτη-μέλη προτού προχωρήσουμε στην κατάθεση μιας νομοθετικής πρότασης από την πλευρά της Κομισιόν. Προφανώς εκεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ε, μεταβατικής περίοδου για τις περιφέρειες αυτές και να είναι ένα σημείο συζήτησης, αλλά το να θεσπίσουμε τώρα μεταβατικές περιόδους και λεπτομέρειες θεωρώ ότι είναι κάπως πρόωρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίλκερ της Κομισιόν. Μας έκανε μια σειρά παρατήρησεων ενδιαφερόντων, ενδιαφερουσών μάλλον, για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και τώρα για να κλείσουμε το θέμα αυτό δίνω το λόγο και πάλι στην κυρία Στάρα Σφεραγκούτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να συνεχίσω λίγο από εκεί που ε, σταμάτησε η Κομισιόν και να συνεχίσω και τις προηγούμενες ε, παρεμβάσεις. Ε, στο θέμα της μείωσης του πληθυσμού μιλήσαμε και με τον ε, εισηγητή της ε, Επιτροπής Γεωργίας. Αυτό δεν, αντικα... δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, αλλά θεωρούμε ότι εμείς αυτό το κριτήριο της μείωσης του πληθυσμού πρέπει να το λάβουμε όταν μιλάμε για τους λεπτούς χειρισμούς. Αν γίνει ο χάρτης, ε, αν γίνει με τα κριτήρια που έχει επισημάνει ε, το Επιστημονικό Συμβούλιο, ε, και κατόπιν γίνεται το θέμα των λεπτών χειρισμών, λαμβάνοντας υπόψη και τον, την απομάκρυνση του πληθυσμού και ε, αυτό δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση Επιτροπή Γεωργία. Για μας είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί. Ε, η τοπική προσαρμογή είναι πολύ σημαντική ε, και η συνεισφορά των κρατών μελών να λάβουμε υπόψη πάντα την πραγματικότητα τη κάθε περιοχή και του κάθε κράτους μέλου. και φυσικά θα πρέπει να δοθεί εκ νέου αξία στις μειονεκτούσε περιοχέ. Τώρα όσον αφορά τις γαλλικές υπερπόντιε περιοχέ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που ισχύει είναι ότι με τα οκτώ επιστημονικά κριτήρια θα γίνει μία νέα προσαρμογή. Δεν ξέρω αν οι υπερπόντες γαλλικές περιοχές βρίσκονται ήδη στον κατάλογο των ε, περιοχών ε, με συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Λογικά θα βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο, στις ορεινές περιοχές, στις ε, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και με ρώτησε και κάποιο αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις ε, περιοχές οι οποίες έχουν ρηπανθεί από χημικούς ε, ρηπαντέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Διερευνητική Ομάδα να λάβει υπόψη μια σειρά από κλιματικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και δημιουργήθηκε μια ομάδα αξιολόγησης. Η ομάδα αξιολόγησης ε, μελέτησε το θέμα του μορφολογία του εδάφους, του κλίματος, ε, ήταν επιστήμονες εγνωσμένου κύριους και ε, συντονίστηκαν οι, οργανι... Ε, οι ομάδες ε, και δημιουργήθηκαν αυτά τα οχτώ επιστημονικά κριτήρια γεωμορφολογικά και κλιματολογικά και λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους ε, παράγοντες ανά την Ευρώπη. θα ληφθεί λοιπόν αυτό υπόψη, αλλά ακούγοντας πάντα και τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα, το πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβατική περίοδος, με ρώτησε κάποιος. Εγώ για τη μεταβατική περίοδο δεν μίλησα, διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί ο χάρτης, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και μετά να γίνει η τελική αξιολόγηση. Και επίσης, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε είναι ευπρόσδεκτο, πιστεύω ότι θα βελτιώσουν ε, το σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ ή τουλάχιστον οι περισσότεροι συμφωνούμε για το θέμα της μείωσης του πληθυσμού και ε, τη συμπερίληψή του στους λεπτούς χειρισμούς. Ευχαριστώ. vielen Dank. Dann... Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο λοιπόν. Οι προθεσμίες για τις τροπολογίες έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9. Είναι η έκθεση, η γνωμοδότηση μάλλον, <clears throat> για το αηφόρο μέλλον για τις μεταφορές με εισηγητή τον κύριο Σιόν Κέλλη, από τον οποίο θα ζητήσω να μας κάνει μια παρουσίαση του ζητήματος αυτού. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή ούτως ή άλλως είναι αργά το απόγευμα, ελπίζω να μην καθυστερήσω. Είναι χαρά μου να είμαι συντάκτης ε, της συγκεκριμένη νομοδότησης. Όλοι γνωρίζετε ότι η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ε, δυνατόν να υπάρχει χωρίς να υπάρχουν ε, οδικά ε, δίκτυα, μεταφορικά δίκτυα. Βέβαια, εάν δεν έχουμε ανταγωνιστικά μεταφορικά μέσα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνιστόσα. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ε, εγώ ζω στην νότια Ιρλανδία, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιφερειάς μου και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι μεταφορές. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα υφόρο μέλος για τις μεταφοράς προς, ε, μια προς έναν ολοκληρωμένο ε, και φιλικό προς το χρήστη σύστημα. Πρόκειται για σχέδια για να βελτιώσουμε τις μεταφορές μας. Ε, θέλουμε να είναι ολοκληρωμένες, να μην είναι διάσπαρτες οι μεταφορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο στις μέρες μας διότι υπάρχει ένα συνεχής αγώνας να έχουμε πιο αποτελεσματική κατανάλωση καυσίμων, ε, να έχουμε καλύτερα, ε, πιο ευέλικτες μεταφορές και όσον αφορά τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι και φιλικές προς το χρήστη οι μεταφορές. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, για την περιφερειακή διάσταση, προσπάθησα να χρησιμοποιήσω ε, τα όσα πολύ καλά έκανε το προηγούμενο, το, η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο και επισημάνθηκε ότι πρέπει να υπάρχουν περιφερειακά αεροδρόμια και να λαμβάνεται υπόψη ε, το θέμα αυτό και να υπάρχουν και προτεραιότητες. Ε, η χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς, ε, καλή σιδηρόδρομη, καλή ναυτιλία και τέλος μια πολύ ειδική μνήμα στις ταχύες σιδηροδρομικές γραμμές. Όσον αφορά στι οδικέ μεταφορέ, θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή κυκλοφορία, κυρίω διαμεθοριακή, και θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσει λοιπόν για να βελτιώσουμε και τη διαμεθοριακή διάσταση των μεταφορών. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που είναι και τεχνική το σύνορο σε κάποιο βαθμό. Να σας παραπέμψω στο 1981, είδαμε τι μειονέκτημα είχαμε τα τελευταία χρόνια ε, και πόσο έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε μια ειρηνευτική διαδικασία και έχουμε πλέον ένα συνειδηρόδρομο που πηγαίνει από το ε, Δουβλίνο στο Μπέλφαστ, ε, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιλλανδίας και θα πρέπει να σκεφτόμαστε γενικώ ολοκληρωμένα. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα είτε σε τοπικό είτε σε οποιαδήποτε άλλο επίπεδο που διότι αν δεν υπάρχουν υποδομές σε τοπικό επίπεδο μπορεί απλώς να, έχουμε, να κυνηγάμε χήμερες και να μην έχουμε αποτελέσματα. Λαμβάνουμε υπόψη και το θέμα των εναέριων μεταφορών κυρίως για τις νησιωτικές και τις ε, εξόχως αποκεντρωμένες περιοχές, τις οποίες επανειλημμένως αναφέραμε σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις κατάλληλες μεταφορές. Το να υπάρχει ένα περιφερειακό αεροδρόμιο σε αυτές τις περιοχές είναι βασική πτυχή για να έχουμε ανάπτυξη. Και στην περιοχή μου, στο Κέρι, ε, η δημιουργία του αεροδρομίου εκεί μας έδωσε τη δυνατότητα διασύνδεσης με το Δουβλίνο, το Λονδίνο ε, και με άλλες περιοχές που καταλαβαίνετε πόσο διευκόλυνε τη ζωή μας οι εξελίξεις στον ενέργειο τομέα τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την απελευθέρωση της αγοράς, ε, βοήθησε ουσιαστικά και όλα αυτά έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους να ταξιδεύουν πολύ περισσότερο. Το μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει τεράστια αύξηση εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Ε, βλέποντας και το 2020 ή και τα επόμενα χρόνια και επομένω όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε είναι να έχουμε έναν πολύ καλά ανεπτυγμένο ε, σιδηροδρομικό τομέα με τρένα ταχείας μεταφοράς και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα πακέτα, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Είδαμε πόση επιτυχία έχουν τρένα όπως το Eurostar, το ταλί βρυξελλες παρισι βρυξελλες αμστερνταμ ε, πολύ γρήγορα τρένα και όλοι οι πολίτες δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει μεγάλη χαρά, ε, διασχίζουν την Ευρώπη με πολύ γρήγορα τρένα και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο μέλλον. Το να χρησιμοποιούμε λοιπόν τέτοια πολύ γρήγορα τρένα ίσως να είναι το μέλλον μας. Εν κατακλείδη να πω ότι η πολιτική συνοχή είναι σαφώς πολύ περισσότερο από καλές μεταφορές, αλλά δεν υπάρχει πραγματική συνοχή χωρίς μεταφορές. Επομένως, η πολιτική συνοχή έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ιστορικά και θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο για το μέλλον. Περιμένω σχόλια από τους συναδέλφους και σαφώς ε, με χαρά θα λάβω υπόψη τα σχόλιά σας και θα συμπεριλάβω στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. <clears throat> Κύριε Κέλλη, έχουμε τώρα διάφορους ομιλητές. Τέσσερις, ο κύριος Κουτμάινης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του εισηγητή μας σε μια σειρά προτάσεων που ίσως θα είχαν ενδιαφέρον για την εκθέση του. Πρώτα απ' όλα, το δεύτερο σημείο των προτάσεών σας. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα θέματα των διασυνοριακών σχεδίων. Τι σημαίνουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα συνδρομικές συνδέσεις οι οποίες συνδέουν χώρες παραγωγός χάρη. Όπως είπε και ο υποψήφιος επίτροπος, η τάση του ήταν να χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία μέσα στις χώρες και όχι τόσο πολύ διαμεθοριακά. Αυτό είναι κρίμα αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία. Δεύτερον, για τα προβλήματα των σιδηροδρόμων. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο πολλές φορές. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει το εισιτήριό του σε ένα επίπεδο πανευρωπαϊκό παραγωγός χάρη όπως το κάνουμε με τις αεροπορικές Μπορούμε εκεί να έχουμε κάποιες προτάσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα σιδηροδρομικά συστήματα. Τρίτο σημείο, όχι μονάχα η ακτοπλοεία, αλλά και οι εσωτερικές, η χρήση εσωτερικών πλοήμων οδών. Υπάρχουν λοιπόν οι δυνατότητες που δίνονται από την αυσιπλοεία σε ποταμούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα μπορούσε λοιπόν να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Χρησιμοποιώντας νέες πράσινες τεχνολογίες. για τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Πρέπει να δώσουμε πάλι έμφαση στο ρόλο των ε, αεροδρομίων. Και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καθαρότητα των ουρανών και της ατμόσφαιρας και πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των εταιριών οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή την ευθύνη των αεροπορικών συγκοινωνιών και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρά το πρόβλημα αυτό της προστασίας του περιβάλλοντο. Αλλά όλα αυτά ίσως θα ήθελα να τα λάβει υπόψη ο εισηγητής και ελπίζω ότι θα μπορούσε να τις υποστηρίξει και αυτές τις προτάσεις και να τις διαβιβάσει και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμμεριστώ τις απόψεις μου με τον εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν μεταφορές σαν εργαλείο εδαφικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής συνοχής. Την ισότητα ελευθεριών επίσης που προωθούν μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την προσέγγιση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών εδαφών που εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες. Και θα ήθελα, όπως προηγουμένως έπραξε και ο κύριος Κέλλη, να τονίσω και τον ρόλο των υπερπεριφερειακών περιοχών, διότι θεωρώ ότι χρειάζεται να υπάρξουν ιδιαίτερες προσπάθειες και μια ιδιαίτερη <clears throat> πολιτική η οποία θα αφορά αυτές τις περιοχές. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε σχέση με τον προλαλήσαντα. ο οποίος μίλησε για κάποια μικρά προβλήματα της πολιτικής των μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο. Νομίζω ότι η περιοχή μας μιλάει ήδη για περιφέρειες και μακροπεριφέρειες και τα διασυνοριακά σχέδια είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι συγκοινωνίες σε όλη την Ευρώπη, οι μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ούλριθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιχειρήσω να επιστήσω την προσοχή του εισηγητού στο εξή. Πριν από μερικούς μήνες δουλεύαμε με την Ετροπή Μεταφορών σχετικά με την αστική κινητικότητα. Έγινε τότε μια μεγάλη, ε, συζήτηση ε, με τα κρατημέλη και κάποια από τα ε, μέλη, δεν ήθελαν ούτε καν ε, να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, λέγοντας ότι αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και μάλιστα των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων ε, βάσει της ε, επικουρικότητας. Στο σημείο 5 υπογραμμίζουμε την ανάγκη εύκολης πρόσβασης αλλά νομίζω ότι σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε τι γίνεται όσον αφορά τα συμπεράσματα ε, της συζήτησης και των εκθέσεων ε, για την αστική κινητικότητα. Γιατί υποτίθεται ότι θα έβγαινε κάτι σαν λευκή βίβλος. Επομένως να ρωτήσουμε τι έγινε με όλο αυτό και να το προσθέσουμε στην παράγραφο 5. Δεν, δεν πρέπει να αναμασούμε απλώς ε, τα πράγματα που έχουμε πει εκατό φορές, ε, ίσως κάτι καινούριο. Αυτό που συζητήθηκε λοιπόν πριν από κάποιους μήνες στο Κοινοβούλιο και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι και βάσει των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί από τη συζήτηση για την αστική κινητικότητα κτλ. κτλ. Ευχαριστώ κύριο Μάια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα είναι ένα φιλόδοξο και καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένε συγκεκριμένε διατυπώσει. Η γνωμοδότηση τονίζει ότι ο στόχος είναι να κινηθεί προς την κατεύθυνση της μελλοντική αηφόρου πολιτικής μεταφορών και μιλάει για υπηρεσίε υψηλή ποιότητα για τους πολίτες στις μεταφορές που πρέπει να ληφθεί υπόψη εκεί και η αρχή της αηφορίας. Εδώ όμως απαιτείται να εξασφαλίσουμε και μία υπηρεσία προς τους πολίτες, δηλαδή εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών αυτών. Να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα είναι αρκετά ελκυστικές και οι δημοτικές υπηρεσίες και ότι δεν θα χρησιμοποιούν μονάχα τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα οι πολίτες. Γιατί δεν έχει επιληθεί το θέμα της μετακίνησης στις, ε, στους Δήμους <clears throat> από τον τόπο εργασίας, στον τόπο ε, διαβίωσης και τούμπαλιν. Όλα αυτά είναι ζητήματα σαφή τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στα πλαίσια των μεταφορών και οδηγούν πάρα πολύ στις κυκλοφοριακές συμφορήσεις πολλές φορές και επομένως και στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Το να μπορέσουμε λοιπόν να περιλάβουμε και αυτή την προβληματική είναι κάτι το οποίο για μένα είναι κάτι επίγον <clears throat> και θα ήθελα αυτή η πρόταση, αυτή η γνωμοδότηση να αναφέρει και το θέμα της αστικής κινητικότητας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνερ. Κυρία Μάνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Σύμφωνα ε, εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις προτάσεις του. Αλλά να πω σύντομα, επί του σημείου 7, όταν γίνεται ε, λόγος ε, στις ε, πιο απομακρυσμένες περιοχές ε, και την πρόσβαση σε αυτές ε, μέσω θαλάσσιων μεταφορών. Βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και οι εσωτερικές πλούτες οδοί είναι επίσης εξίσου σημαντικές ε, και εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε και στις λίμνες. Ε, θα ήθελα στο τελικό σχέδιο να υπάρχει αναφορά και στις λίμνες. Als Ευχαριστώ. Η κυρία Ντέιλι, η τελευταίος ομιλητής μας. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Κέλλη για την ε, ε, έκθεσή σας την γνωμοδότηση αυτή, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Μετά την αποτυχία της Κοπενχάγης, η γνωμοδότηση αυτή μας δίνει τροφή προσκέψη και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την πολιτική των μεταφορών με τρόπο συνολικό. Νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τους σιδηροδρόμους έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω χρηματοδότηση των, χερσαίων, υποδομών χερσαίων μεταφορών ε, εκτός από ειδικέ περιπτώσεις. Τέλος, στις πόλεις θα πρέπει να ε, ε, κάνουμε καλύτερες τις δημόσιες συγκοινωνίες, κυρίως δε ε, να έχουν πρόσβαση καλύτερες σε αυτές οι λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές και επίσης να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η οικοδόμηση αυτών των περιαστικών περιοχών στις μεγάλες Μητροπόλεις. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ε, ενθαρρύνουμε τις ε, μεταφορές μικρών αποστάσεων και να αποκεντρώσουμε επίσης και να αποδυναμώσουμε τα μεγάλα λιμάνια. Άκουσαμε πολλές εκκλήσεις υπέρ των σιδεοδρόμων. Πριν από τον εισηγητή θα ήθελα και πάλι να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Σαντανάφο ή κάπως έτσι, συγγνώμη που κακοποιώ το όνομά σας. Well, Μπορώ να σας πω <clears throat> ότι πολλά από τα σχόλια τα οποία έγιναν εδώ αναφέρονται σε ζητήματα τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την συνέχεια που θα δοθεί στην εργασία μας για το μέλλον των μεταφορών, στην ανακοίνωση λοιπόν αυτή της Κομισιόν, η οποία είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια νέα λευκή βίβλο για τις μεταφορές, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί στο τέλος του επόμενου χρόνου, του τρέχοντος χρόνου μάλλον, ή στις αρχές του 2011. Από αυτή την έννοια, αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να τη δούμε σε αυτό το φως και θα λάβουμε υπόψη και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία του λευκού αυτού βιβλίου. Ευχαριστούμε για την, την παρατήρηση της Κομισιόν και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κέλλη, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις που μου έκαναν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Ε, χαίρομαι που άκουσα ταύτιση απόψεων όσον αφορά τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, ε, όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και επίσης ότι θα πρέπει να βρεθούν φιλικοί προς τον χρήστη μέθοδοι ας πούμε για να βγάζει κανείς τα εισιτήριά του ή να κάνει τις κρατήσεις του κτλ. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα και βεβαίως και όλα αυτά που είπατε σχετικά με τις low cost εταιρείε, Ryanair κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όσον αφορά τώρα τις θαλάσσιες μεταφορές, βεβαίως και οι εσωτερικές πλωτές οδοί είναι πολύ σημαντικές. Η εσωτερική ναυσιπλοεία, ας πούμε, ε, ε όπως είπατε, ε, λίμνες και ποτάμια, βεβαίως θα ληφθεί υπόψη και αυτό. Ε, η σχέση ανάμεσα στις καθαρότερες μεταφορές, τον καθαρότερο ουρανό, καθαρότερη ατμόσφαιρα, κλιματικές αλλαγές, η σχέση είναι πάρα πολύ στενή ασθενή και βεβαίως εναλλακτικές ε, ε, λύσεις ε, είναι ευπρόσδεκτες. Τώρα πιστεύω ότι η συμβολή όλων ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική, είτε έγινε αναφορά στην αστική κινητικότητα και τη συζήτηση που είχε γίνει τότε για το θέμα αυτό, ε, είτε ε, ανεφέρθη η καλύτερη αντιμετώπιση των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαίρομαι που ε, όλοι οι συνάδελφοι διάβασαν την έκθεση και προσπάθησαν να συμβάλλουν ε, σε αυτήν, ε, γιατί ούτως ή άλλω η αλλω η εκθεση θα αντικατοπτρίζει τις συλλογικε σκέψεις αυτής της Επιτροπής και βεβαιω θα ληφθούν υπόψη οι απόψη όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω, έχω να κάνω κάποια παρατήρηση. Απλώς εγώ θα ήθελα να πω ότι καμία οδική μεταφορά δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά όσο η καλύτερη σιδηρόδρομη. Έρχομαι τώρα στην ε, προθεσμία τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 22 Φεβρουαρίου. Κλείνει λοιπόν το σημείο αυτό της ημέρησης διάταξης. Περνάμε στο επόμενο. για την τροποποίηση του κανονισμού 247 του 2006 για τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Τισιέρα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα όσο το δυνατόν πιο σύντομα να συμμεριστώ ορισμένες βασικές ιδέες, τις κομβικές κατά κάποιο τρόπο ιδέες της Κομισιόν σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού 246 του 2006 που θεσπίζει μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό ακολουθεί το αντίστοιχο άρθρο τη ε, Συνδίκη Λισαβόνα. που λέει ότι οι περιοχέ αυτές οι οποίες έχουν μόνιμα μειονεκτήματα λόγω παραδείγματο χάρη γεωγραφικής ε, θέσης, μικρής, ε, μικρής επιφάνειας, νησιωτικού χαρακτήρα και περιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ότι πρέπει να καλύπτονται στο πλαίσιο αυτό. Όλοι μας θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η ρήτρε αυτού του κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαίτερε καταστάσει σε αυτέ τι περιοχέ και στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να αντανακλούν και την εξέλιξη των τοπικών αγορών. Εξάλλου αυτά τα μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερε τρευλώσει αγορά, γιατί τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίε παράγονται και καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο. Λόγω της τεχνικότητας αυτού του θέματος θα σταθώ μονάχα σε μερικά βασικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές εγώ μπορώ να υποστηρίξω πλήρως την πρόταση της Κομισιόν, ιδίως σε τρία θε... κομβικά σημεία, σημαντικά σημεία. Κατά τη δυνατότητα στις Αζόρες να υπάρχει εισαγωγή του ακατέργαστου ζαχαροκάλαμου μέσα στις δυνατότητες παραγωγής στα Κανάρια να μπορούν να, μπορούν να συνεχίζουν να εισάγουν γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή του πληθυσμού εκεί και στις, ε, στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα να υπάρχει παραγωγή γάλακτος για τοπική κατανάλωση. Αλλά, <clears throat> καταρχήν, μέσα στις τροπολογίες μου υπάρχει μια πρώτη ομάδα έξι τροπολογιών που θέλω να συζητήσω και με τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους αφορούν το εξή θέμα. Δύο από τις τροπολογίες αφορούν την πρόταση της Κομισιόν και τέσσερις έχουν να κάνουν με το αρχικό κείμενο του κανονισμού. Η πρώτη θέλει να άρει την ασυμμετρική μεταχείριση των αζωρών έναντι της Μαδέρας και επίσης το, τη μεταχείριση των δύο αυτών περιοχών σε σχέση με ορισμένε καλλιέργειες οι οποίες δεν επιτρέπεται να ε, να γίνονται στις συνθήκες αυτές. Επίσης, σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση των αγροτικών αγορών, υπάρχουν συγκεκριμένες μνήες και ρυθμίσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Η δεύτερη τροπολογία έχει να κάνει με τον αναδρομικό χαρακτήρα της εφαρμογής αυτού του κανονισμού και η τρίτη τροπολογία έχει σαν στόχο να διευκρινίσει καλύτερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η παραγωγή μεταποιημένων και μη μεταποιημένων προϊόντων που έχουν τύχει τέτοια επιδότηση και υποστήριξη από αυτό το καθεστώ μπορούν να τύχουν εξαγωγή. Αυτή η τροπολογία, όπω και η τέταρτη και πέμπτη τροπολογία, έχουν σε στόχο να βελτιώσουν την ευκαμψία στα κράτη-μέλη από τα οποία γίνεται η τροφοδοσία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες των υπερπεριφερειακών περιοχών και ο εφοδιασμός των τοπικών αγορών. Το σύνολο αυτών των τριών τροπολογιών προτείνει να υπάρξει τακτική ενημέρωση των ποσοστών, των ποσοτήτων προϊόντων που μπορούν να εξάγονται προς τα υπερπεριφερειακά αυτά μέρη βάσει αυτού του καθεστώτος. Αυτές οι ποσότητες λοιπόν θα πρέπει να καθοριστούν σε σχέση με το μέσο όρο των ε, εξαγωγών των ποσών των ποσοτήτων του 1990-1991, έτσι αποκρισταλώνεται το ιστορικό ο ιστορικός χαρακτήρας αυτών των ποσοτήτων και με τον τρόπο αυτό δεν συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Οι οδηγίες αυτές αναφέρουν ότι τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς τροφοδοσίας θα πρέπει να προταθούν από τις ίδιες τις περιοχές αυτές, τις υπερπεριφερειακές. Πράγματι, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί <clears throat> στη διάρκεια του χρόνου και η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του κανονισμού 247 2006 ανοίγει το δρόμο για την τροποποίηση και άλλων συναφών ε, κανονισμών, όπως 723 του 2006, ο οποίος θεσπίζει ορισμένες ρήτρε και ο οποίος θα πρέπει να τροποποιηθεί σε σχέση με τις μέγιστες ποσότητες εξαγωγής ορισμένων προϊόντων, τα οποία προέρχονται από ειδικά καθεστώτα για τις περιοχές αυτές. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη είναι η μείωση του, της προθεσμίας από 90 σε 30 μέρες για την καταβολή των ε, ποσών αυτών της ε, αρρωγής βάσει και της οδηγίας για τη λεγόμενη ε, καθυστέρηση καταβολής των ε, ποσών αυτών, των αρρωγών και πιστεύω ότι είμαι απόλυτα στη διάθεση των συναδέλφων για να συζητήσω αυτή την ε, γνωμοδότηση, τις δικές μου τροπολογίες και οποιασδήποτε άλλες τροπολογίες θέλετε εσείς θέση. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Κύριος Όγο έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τα λεγόμενα του εισηγητού όσον αφορά τη ζάχαρη για τις αζόρες, καθώς επίσης και για τα γαλακ... προϊόντα γαλάκτος ε, για τα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τώρα για την Ρεϊνιόν, κατανοώ βεβαίως τις καλές προθέσεις ε, του ε, εισηγητού και ως εκπρόσωπος της Ρεϊνιόν θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Όμως, θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ε, στόχο και την προέλευση αυτού του αιτήματος, γιατί μου είπαν ότι μετά από μια επιδημία διαπιστώσαμε ότι ε, χάθηκαν χίλιες γαλακτοφόρες αγελάδες. Όμως φαίνεται ότι παραδόξως δεν μειώθηκε καθόλου η μείωση φρέσκου γάλακτος, η παραγωγή συγγνώμη, φρέσκου γάλακτος και επομένως κάτι συμβαίνει όσον αφορά το, την παραγωγή όσον αφορά μάλλον καλύτερα ε, το, τον καθορισμό συσχετισμού παραγωγής φρέσκου γάλακτος ε, με, γάλακτος, με γάλα σε σκόνη και φοβούμε ότι εάν το καθεστώς ε, της, ε, των ε, Καναρίων επεκταθεί και στην νήσο της Ρεϊνιό, φοβούμε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο ασαφής και επομένως θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται είτε από την κυβέρνηση της Γαλλίας είτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ρεϊνιό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα περαιτέρω αποσαφήνιση ε, των όρων τοπικής παραγωγής. Είναι γεγονός ότι, ότι η ανάγκη ε, γάλακτος και ε, προϊόντων γάλακτος στην Ρεϊνιόν δεν καλύπτονται από την τόπια παραγωγή. Παρόλα αυτά θα ήθελα κάποιες περαιτέρω αποσαφηνείς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες κύριε Πρόεδρε. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τυρολίν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ ε, ε, την εξαιρετική εργασία του κυρίου Τεξέιρα. Και όταν αναφέρεται στην αρχή της επικουρικότητας ε, συμφωνώ απολύτως μαζί του, σε σχέση δηλαδή με τις ε, άκρος ε, περιφερειακές περιοχές και βεβαίως συμφωνώ μαζί του να αναφέρεται στην ανάγκη καλύτερης προσαρμογής των περιοχών αυτών στις ανάγκες της αγοράς έτσι ώστε να υπάρξουν οι βέλτιστες ικανές συνθήκες. Στο αρχικό κείμενο προβλέπει τροποποίηση της ε, παραγράφου 41 του αρχικού κανονισμού που αφορά μονάχα την ε, ε, μαδέρα για τις περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά άκρος περιφερειακές. Τώρα, η δυνατότητα δημιουργίας, ε, η εξαίρεση για την Ρουινιό όσον αφορά τη δυνατότητα ε, δημιουργίας γαλακτοκομικών προϊόντων από γάλα σε σκόνη ε, εισαγμένο από κοινοτικέ χώρες, βεβαίως είναι σωστή και θεμητή για την Ρουινιό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τα άλλα υπερπόντια διαμερίσματα να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Γι' αυτό σας ζητώ ε, να ε, ενταχθεί η τροπολογία κατά αυτή την έννοια στην γνωμοδότηση του συναδέλφου μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέζε ή κάπως έτσι, συγγνώμη δεν είμαι πολύ καλός στην προφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κρέζε λέγομαι. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία φύγονται στην έκθεση αυτή. Το ζαχαροκάλαμο και, η... το γάλα. Εγώ συμμερίζομαι το μεγαλύτερο μέρος των συστάσεων που περιέχονται σε αυτή την έκθεση και φυσικά δεν θέλω να υποστηρίξω την κρίζωση των αμπελιών σε αυτές τις περιοχές. Αλλά θέλω να τονίσω το θέμα της προσαρμογής λόγω κλιματικής αλλαγής που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική μνήμα για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τις περιοχές τις ακροσπεριφερειακές και εγώ δεν καταλαβαίνω τη λογική της ε, απόσταξης λόγω κρίσης γιατί να ισχύει αυτή για τα Κανάρια και όχι για Αζόρες, Μαδέρα και άλλα, ε, άλλα μέρη. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του ζαχαροκάλαμου. Εγώ θα είχα την τάση να υποστηρίξω την έκθεση αυτή και τη ρύθμιση η οποία μας αναφέρεται. Θα ήθελα όμως προηγουμένως να έχω και κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με το από πού θα γίνει η εισαγωγή του ακατέργαστου ζαχαροκάλαμου όπως αναφέρεται. Θα έρθει μονάχα από άλλες υπερπεριφερειακές περιοχές και στην περίπτωση αυτή ποια είναι η άποψη της Κομισιόν σε σχέση με τη δυνατότητα να προέλθει από τις χώρες ΑΚΕ. Για το γάλα. Επανέρχομαι στον κύριο Ορό και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Είμαστε σίγουροι καταρχήν ότι η παραγωγή είναι τόσο λίγη που δεν μπορούμε να έχουμε επάρκεια στο θέμα της γαλακτοκομικής παραγωγής. Δεύτερον, πώς θα προστατευτούν οι μικροί παραγωγοί από τη στιγμή που θα ανοίξει η αγορά για την εισαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος. Και τρίτον, μήπως θα έπρεπε <clears throat> να βοηθήσουμε τους μικρούς παραγωγούς με μια αρρωγή για την ανάπτυξη και όχι να καταφύγουμε στην εισαγωγή γάλακτος σκόνη από, άλλα, από άλλες περιοχές. Είναι μια συζήτηση η οποία είναι λιγότερο τεχνική πιστεύω από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, <clears throat> πραγματικά τελευταίος ομιλητής τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να εκφραστώ σε σχέση με αυτό το σχέδιο αργών που αφορά τον αγροτικό τομέα, νομίζω ότι αυτά που είπε ο και τα συμπλήρωσαν και οι συνάδελφοι, αντανακλά μια αξιολόγηση που πρέπει να γίνει με τρόπο ιδιαίτερα ειδικό για κάθε συγκεκριμένη περιοχή υπερπεριφερειακή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καλλιέργειες που γίνονται σε αυτές τις περιοχές. Επομένως υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη <clears throat> να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την προβληματική που αφορά στις υπερπεριφερειακές περιοχές. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι και κάπως κατεπήγον όπως έχουν τονίσει χώρες και περιφέρειες για την εφαρμογή αυτών των μέτρων και επίσης να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία σε σχέση με τις ε, διαφορές που μπορούν να προέλθουν μεταξύ ημών και της Επιτροπής Γεωργίας, με το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία της συναπόφασης προς ικανοποίηση όλων και ιδίως των υπερπεριφερειακών περιοχών, των άκρως περιφερειακών περιοχών που είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενες και αυτά ήθελα να καταθέσω εδώ. Εντάξει. <clears throat> Τελευταίος ομιλητής ήταν αυτός από τους συναδέλφους. Η κυρία Ιμπέριο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή για τις προτάσεις που ακούστηκαν στην ε, συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση της γνωμοδότησης την οποία διάβασα με μεγάλη προσοχή. Σημειώνομαι ότι κάποιες από τις προτάσεις ε, της ε, πρώτης νομοδότησης ε, προχωρούν πέραν των προτάσεων ε, που συζητώνται και που έχουν προταθεί και επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως είπε και ο κ. Άλβες, νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι μάλλον επίγουσα, είναι μάλλον επίγον το θέμα, γιατί υπάρχουν πρόνοιες οι οποίες αναφαίνονται ε, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν την ε, ανακοίνωση και οι οποίες αφορούν ε, ανταπόκριση σε αίτημα που λάβαμε από τις εν λόγω περιφέρειας. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ήδη την επανεγγραφή της εν λόγω οδηγίας βάσει των νέων στοιχείων και σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως ε, θα ακούσουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις σας έτσι ώστε ενδεχομένως να τροποποιηθούν κατά αυτή την έννοια οι πρόνοιες του εγγράφου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια που άκουσα από τα μέλη της Επιτροπής. Ας πούμε, το γάλα στη σκόνη, το οποίο επιτρέπει πετέ ε, στην Ρεϊνιόν να ε, το εισάγει έτσι ώστε να το κάνει ε, φρέσκο γάλα προς κατανάλωση είναι γεγονός ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τις άλλες για τα άλλα υπερπόντια διαμερίσματα. Αλλά εδώ δεν είναι κάτι καινούριο. Ξέρουμε ότι αυτό το είδους η ανασύσταση και κατανάλωση ε, ανασταθέντος γάλακτος ε, προβλέπεται για τις περιοχές αυτές. Όμως ε, είναι γεγονός ότι τα συγκεκριμένα νησιά, η Μαδέρα δηλαδή και η Ρεουνιόν, ε, λόγω ακριβώς ε, του, του ειδικού γεωγραφικού ανακλήφου, έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη δυσκολία στο να παράγουν την ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς περίπου 20% ε, καλύπτει η τοπική παραγωγή, καλύπτει την ε, τοπική ανάγκη κατανάλωσης ε, και επομένως η Μαδέρα και η Ρεουνιόν υποχρεούνται να εισάγουν ποσότητες γάλακτος σκόνη που ανασυντίθεται επί τόπου στην ε, Γουαδελούπη και την Μαρτινίκα τώρα. Όσον αφορά ε, την, ε, τα νησιά αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε ότι υπήρχε λόγος να επεκτείνει την εξαίρεση και στα δύο αυτά νησιά, διότι το αίτημα το οποίο έλαβε αφορούσε μονάχα και ξεκινούσε μονάχα από την Ρεουνιόν. Όσον αφορά τώρα τα Κανάρια νησιά, εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν περιέχονται στο παράρτημα 1 της ε, συνθήκης και επομένως χρειάζεται ειδική εξαίρεση. Πρόκειται για προϊόν το οποίο είναι αρκετά φτηνό και το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιείται από τα χαμηλά οικονομικά στρώματα του νησιού. Να πω εν παρόδο ότι η Ισπανία ζήτησε να μην υπάρχει χρονικό ε, περιθώριο ε, και ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου αυτό το αίτημα που υπέβαλε η Ισπανία. Όσον αφορά τώρα το κρασί, θα σημειώσω τις παρατηρήσεις τις οποίες άκουσα εδώ και επί των οποίων δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γενικώ θα λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε και αν είναι δυνατόν θα τα συμπεριλάβουμε στην νέα ε, ε, εκδοχή ε, την οποία θα έχετε στα χέρια σας τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2010. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Τισιέρα να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομο στην απάντησή του στα πολλαπλά αυτά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνοπτικά. Έχω καταγράψει όλα τα σχόλια των συναδέλφων, τους οποίους θέλω φυσικά να ευχαριστήσω κιόλα. Απλώς θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσω να εμβαθύνω στο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Σωρό για την Ρέινιόν και το Γάλα. στην περίπτωση της Μαδέρας γνωρίζω ότι ό,τι παράγεται εκεί δεν είναι επαρκές για να καλύψει την ε, εντόπια ζήτηση. Γι' αυτό το θέμα αυτό της ανασύστασης του γάλακτος σε σκόνη ετέθη πρώτα στη Μαδέρα και μετά μεταφέρθηκε στην Ρεϊουνιόν αυτή η προβληματική. Τα υπόλοιπα θέματα επίσης θα προσπαθήσω να τα αντιμετωπίσω μαζί με τους συναδέλφους και στη συνέχεια τα θέσω μέσα στο σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. herzlichen Dank für die... Ευχαριστώ πολύ για την πραγματιστική σα ε, αντιμετώπιση. Θέλω να σας αναφέρω ότι η προθεσμία για τι τροπολογίε και σε αυτή την περίπτωση είναι η 2 Φεβρουαρίου και ότι στις 22 Φεβρουαρίου θα προχωρήσουμε στην, ψηφο, στην ψηφοφορία επί της γνωμοδοτήσεως αυτής. Τελευταίο και λουκούμιο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι νέες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βλασάκ. Ε, κύριε Περσίρη, δημόσιες συμβάσεις ε, όχι μόνο είναι πολύ σημαντικές, αλλά είναι και ε, μία από τις πιο σημαντικές ε, πτυχές, αν δούμε τα θέματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη σήμερα. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, διότι αφορά το 16% όλου του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτό είναι ο όγκος της χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές ε, για να ε, διορθώσουν δρόμους, να αγοράσουν ε, λεωφορεία μαζικής μεταφοράς για τους Δήμους, αλλά και για νοσοκομεία ή γραφεία. Η Επιτροπή μας ασχολείται με το θέμα των δημόσιων συμβάσεων από πλευράς της εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και όσον αφορά και στον τελικό ε, χρήστη, τους δήμους, τους πολίτες, τις κοινότητες. Οι δημόσιες συμβάσεις ε, στα προγράμματα τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένες φορές ε, δεν ε, αποτελούν και ιδιαίτερα επιτυχές αντικείμενο. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από το ελεγκτικό συνέδριο τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι τα θέματα δημόσιων συμβάσεων είναι από τα πιο επικίνδυνα όταν υλοποιούνται έργα τα οποία έχουν ε, ε, χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που διαπιστώνουμε συνήθως είναι παραβίαση των όρων του σύμβασης, ε, λάθη στην τεκμηρίωση ή και κάποιες τυπικές ελλείψεις συχνά το πρόβλημα δεν είναι τόσο η παραβίαση κάποιου κανόνα όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αλλά κυρίως το θέμα της εφαρμογής. Ε, οι διαχειριστές αλλά και οι πόλεις ή οι δήμοι πολύ συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες νομικές γνώψεις, δεν έχουν την ανάλογη κατάρτιση και δεν κατανοούν πολύ καλά τους κανόνες που βρίσκονται στη βάση των δημοσίων συμβάσεων. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τους κανόνες που διέπουν τέτοιες συμβάσεις, σίγουρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαι πεπισμένος ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προάγουν την ε, κατάλληλη επιμόρφωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να περιπλέξουμε τις αρχές και τους όρους μιας διαδικασίας που είναι αφεαυτές ιδιαίτερα περίπλοκη. Υπάρχει και μια κάποια έλλειψη διαφάνειας. Και υπάρχει και μεγάλη γραφειοκρατία. Ορισμένες φορές είναι τεράστιε οι δραστηριότητε, οι διαφορές μεταξύ συμβάσεων και δραστηριοτήτων στις δημόσιες συμβάσει. Υπάρχει και το τι γίνεται στην περίπτωση της απόφασης ε, να γίνουν ε, δημόσιες συμβάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν και προβλήματα στις ε, ε συμβάσεις ιδιωτικού δημοσίου και όλα αυτά φυσικά αποτελούν προσκόμματα διότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί κανόνες και εδώ είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποιες αλλαγές. Κατά την ε, πρόταση λοιπόν, την εκπόνηση αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης χρησιμοποίησα τις ε, απόψεις ενδιαφερόμενων φορείων όπως του Eurocities και χρησιμοποίησα τις γνωμοδοτήσεις τους και είδα και κάποια πιο συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ε, μπορεί να προκύψουν στο θέμα των δημόσιων συμβάσεων. να ευχαριστήσω και τους ε, εταίρους για τη συνεισφορά τους. Τα έχω συμπεριλάβει και στη γνωμοδότησή μας κάποια στοιχεία. Και να σας πω ότι συζήτησα την πρόταση και με την επί της ουσίας ε, αρμόδια εισηγήτρια την Επιτροπή ΙΜΚΟ, την Χάιντε Ρούλε, η οποία είναι παρούσα σήμερα εδώ και με τη Σαμπίνε Χάιον και τον Πίτερ Σίμονς με τους συναδέλφους καταλήξαμε σε μια συμφωνία και θεωρούμε ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί. Η αρχή της αυτοδιαχείρισης, μια κάποια ελευθερία σε θέματα συνεργασίας είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής επικουρικότητας και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν προβλήματα, διότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι πολύ σαφής και σε κάποιες περιπτώσεις ε, είναι πολύ αυστηρή στα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή όλο το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί σαφώ θα αυξηθεί το γραφειοκρατικό άγχος. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ενδιαφέρον και να εφαρμόσουμε με τον κατάλληλο τρόπο τις νομικές ρήτρε που ήδη ισχύουν. Ε, θα ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την κατεύθυνση με τους συναδέλφους για να δούμε πώς μπορούμε να διατυπώσουμε με τον σωστότερο τρόπο τα όσα παρουσιάζονται στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τρεις ομιλητές και σας παρακαλώ, τέσσερις μάλλον, σας παρακαλώ να είστε σχετικά σύντομοι λόγω του χρόνου. Ο κύριος Σίμων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάζακ για αυτό το πρώτο σχέδιο, για το ανοιχτό πνεύμα και τη διαθεσιμότητά του να συνεργαστεί μαζί μας και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση συνολική που να είναι ικανοποιητική για όλους μας. Τρεις παρατηρήσεις θα επιτρέψω στον εαυτό μου σήμερα. Η πρώτη σε σχέση με την συνεργασία μεταξύ Δήμων. Στο σχέδιο του κυρίου Φλάσακ η συνεργασία των Δήμων αυτών την έχει τονίσει ο κύριος Βλάσακ, έχει τονίσει την ανάγκη να υπάρξουν ε, βιώσιμα σχέδια για την υδροδότηση και την αποχέτευση και η σημασία φυσικά στον τομέα αυτό είναι όλο και μεγαλύτερη. Υπήρξε θετική νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 2007 για το θέμα αυτό, την οποία εμεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νομολογία πράγματι γίνεται κομμάτι τη καθημερινή πρακτική τη Κομισιόν χωρί καμία απολύτω εξαίρεση. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το σημείο 4 του σχεδίου γνωμοδότηση του κ. Φλάσακ, ο οποίο αναφέρθηκε στην εταιρική σχέση μεταξύ των φορέων αυτών. Πρέπει να είμαστε εδώ σαφείς στο σημείο αυτό. Η γερμανική μετάφραση για μένα είναι τελείως λανθασμένη, ίσως πρέπει να ελέγξουμε και άλλες γλωσσικές μορφές. Λέει ότι όταν υπάρχουν PPP, οι λεγόμενες PPP, οι Public-Private ε, Partnerships, <clears throat> ενώ στη συνέχεια το γερμανικό κείμενο δεν αναφέρεται σε εταιρικέ σχέσει δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, αλλά σε διαδικασίε για τι δημόσιε προμήθειε, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια ε, διόρθωση των κειμένων και αυτό να ληφθεί υπόψη και στην ε, πρόθεσμη για τις τροπολογίες. Πάντως, πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις και οι προτάσεις για τις συνεργασίες δημοτικού και ιδιωτικού τομέα μέχρι στιγμής δεν έχουν επιφέρει καμία απλοποίηση στην περίπτωση των προμηθειών και έχουν φέρει μάλλον περισσότερη ανασφάλεια δικαίου. Κάτι ακόμα το οποίο θα να τονίσω αφορά <clears throat> τις προηγούμενες περιπτώσεις, τις παλιές περιπτώσεις, τις ιστορικές περιπτώσεις, οι οποίες προέρχονται από στιγμές πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η Γενική Εισηγήτρια του Δικαστηρίου δεν μπόρεσε, δεν, έχει μια πρόταση για αυτές τις παλιές συμβάσεις που υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο εμεί θα εγγράψουμε στο νέο νομικό πλαίσιο αυτές τις ε, ιστορικές συμβάσεις. Έρχομαι και πάλι στο σημείο 6 του κυρίου Φλάσακ. Εδώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δούμε για μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μια <clears throat> ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε τις προδιαγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες στην περίπτωση που εμπλέκεται ο δημόσιος τομέας. Χαίρομαι που λαμβάνετε υπόψη την ε, αρχή της επικουρικότητας και προχωρώ στον κύριο Ματούρα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι πολύ που έφτασε στα χέρια μας αυτή η πρόταση που συζητούμε σήμερα. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι όταν αναφερόμαστε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να ομολογήσουμε ότι στον τομέα αυτό αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα και αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εξελίξει όσον αφορά τους ε, κανόνες που θα διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και το νομικό πλαίσιο, γιατί έτσι θα μειωθούν οι κίνδυνοι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα ε, όσον αφορά την χρήση των διαρχοτικών ταμείων. Το λέω αυτό γιατί η έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου οδήγησε σε προβλήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση νομοθεσίας την εθνική νομοθεσία. Και μερικές φορές ε, η κατάσταση ε, περιεπλάκει ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες. Παράδειγμα, η Ρουμανία πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και τώρα, έχει προβλήματα με ε, τις περιόδους που αναφέρονται στις διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Μερικές φορές το, το χρονικό διάστημα είναι τεράστιο. Ε, πολλές φορές χρειάζεται να περιμένει κανείς χρόνια μέχρι ότου έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Επομένως, αυτού του είδους το νομικό πλαίσιο σημαίνει ότι εμείς χάνουμε διαρκώς κονδύλια. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερως που απλουστεύουν οι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάτρο. Κυρία Φερχάιμ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάσεκ για το σχέδιο αυτογνωμοδότηση και φυσικά και για την πολύ καλή συνεργασία που είχε με όλους μας ήδη προηγουμένως. Έχει τονίσει μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία και το νομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις δημόσιες ε, συμβάσεις έχει γίνει σαφές μετά από το 2004 Έχουμε πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει ερμηνεύσει τα σημεία όπου υπήρχε ακόμα ασάφεια και έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα είναι διαφάνεια στην μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή στις ε, συγκεκριμένες χώρες και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση σε σχέση με τις συμβάσεις. Εγώ χαίρομαι ότι ο κύριος Βλάσεκ τόνισε ιδιαίτερα την απαραίτητη περισσότερη κατάρτιση, περισσότερη πληροφόρηση <clears throat> για τα διάφορα επίπεδα, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Αυτό φυσικά είναι καθήκον των εθνικών κρατών που έχουν το καθήκον, έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εθνικό επίπεδο και από την άποψη αυτή, όπως είπε και ο κύριος Ματούλα, είναι φανερό ότι κάποια κράτη έχουν προχωρήσει περισσότερα από τα άλλα και κάποια κράτη είχαν μεγάλες δυσκολίες στην περίπτωση των διαφθορτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι αυτή η γνωμοδότηση και οποιαδήποτε έκθεση πρωτοβουλίας δεν νομίζω ότι θα διαλάβει το θέμα της αλλαγής του νομικού πλαισίου. Απλώς πρόκειται για την ανάγκη να έχουμε μια πιο διάφανη δομή εφαρμογής αυτών των μέτρων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία τονίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος των Δήμων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών βάσει και της συνθήκης Λισαβόνας που έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και επίσης τονίζεται η αρχή της ε, επικουρικότητα, ότι θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται σε <clears throat> όλες αυτές τις αντίστοιχες δομές ή επίσης στην περίπτωση εκχώρησης εξουσιών. Θα πρέπει να παραμείνουν λοιπόν οι εξουσίες καταρχήν στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ό,τι αφορά την, ε, σύμβαση για παροχές υπηρεσιών βάσει και τις οδηγίες για τις υπηρεσίες και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε επίπεδο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, να διατηρηθεί λοιπόν στα πλαίσια της επικουρικότητας η απαραίτητη ευελιξία και ελευθερία που έχουν αυτοί οι φορείς για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Φεράιν. Ο κύριος Γκουτμάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις πολύ επαγγελματικέ προτάσεις σας, τολμώ να πω, και συμφωνώ ότι το πρώτο και το πιο βασικό είναι αυτό που α, διάβασα στην έκθεση. Τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση αυτών των διαδικασιών. Γιατί αυτό, διότι αν δείτε το νέο πρόγραμμα, το Urban, το οποίο εφαρμόζεται ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, θα δείτε πάρα πολύ εύκολα ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν είναι και τόσο καλή στα εθνικά προγράμματα που σημαίνει ότι τα urban, τα οποία είναι αστικά προγράμματα, δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί το πρόβλημα να είναι η συνεργασία και η υποστήριξη υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο που είναι υπεύθυνε για την διαχείριση των κονδυλίων και ε, τη διαχείριση των τοπικών αρχών να πω ότι δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στα παλιά κράτη-μέλη, αλλά στα νέα κράτη-μέλη έχω κάποια πείρα. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία εκπονήθηκαν πάρα πολύ καλά, μεν, αλλά στην πράξη δεν λειτουργούν καθόλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων, μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη εμπιστοσύνης, διότι η σχέση μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο των αρχών, απέτυχαν. Και δεν ξέρω κατά πόσον ε, αυτό είναι νέα νομοθεσία, είναι κάτι άλλο που χρειαζόμαστε, αλλά υπάρχει ανάγκη να δούμε τι γίνεται με προγράμματα όπως τα PPP, τα οποία δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Jan Olbrecht και μετά ο Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Ένα γιατί μάλλον υπάρχει κάποια παρανόηση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα Urban. Αυτά τα προγράμματα τελειώσανε το 2006. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι κάποια προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τις πόλεις, αλλά το Urban δεν υπάρχει πια. Ήταν στο Disability 2006. Σύμφωνα με, δεύτερο στοιχείο, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, ε, ένα από τα κυριότερα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε λάθη ε, είναι οι, δημόσιες, ε, οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε όλα τα επίπεδα και τοπικά και περιφερειακά. Νομίζω λοιπόν ότι το ερώτημα είναι εάν όλα είναι σαφή από πού προέρχονται τα λάθη, άρα πού είναι το πραγματικό πρόβλημα και γιατί έχουμε συνέχεια τόσα πολλά λάθη όσον αφορά την πρόσκληση υποβολή ε, προσφορών στις, ε, στους δημόσιους Θα προσπαθήσει τώρα ο εισηγητή να απαντήσει στο ερώτημα αυτό και πάλι θα δώσουμε το ρόλο στην Κομισιόν και μετά ο κύριος Βλάσακ. Η κυρία, η κυρία, η κυρία εισηγήτρια, εγώ ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που μου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστώ. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το ρόλο του κ. Βλάσακ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά. Να έρθω τώρα στα θέματα τα ουσιαστικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί τώρα όλα αυτά τα θέματα των δημοσίων συμβάσεων ως, ως μια εργαλειοθήκη για πάρα πολλά θέματα. Εγώ ως πράσινη θα ήθελα αυτά να χρησιμοποιηθούν και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και στην, στον τομέα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μορφή συντονισμού σε σχέση με όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίε γίνονται. Εγώ πέρασα μια μέρα ψάχνοντας στο ίντερνετ για να καταλάβω τι γίνεται για τα θέματα αυτά της, ε, ε, των δημοσίων προμηθειών. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοδήποτε Δήμος να ελέγξει όλες αυτές τις προδιαγραφές που βρίσκονται δεξιά και αριστερά, τους κανόνες προτού προχωρήσει στη σύναψη μιας σύμβασης. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει ένα ιδιαίτερο ρόλο στις ε, κοινότητες, τους δήμους, τις περιφέρειες <clears throat> για να φέρουν σε πέρα σε αυτό το έργο είναι απαραίτητο να υπάρξει η εκπαίδευση, η τεχνική βοήθεια αλλά δεν θέλουμε να πάρει μια μορφή ήπιου νόμου μέσα εισαγωγικά και να υπάρχει μια πολυπικιλία προσεγγίσεων για το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να υπάρξει και υπερβολικός φόρτος γραφειοκρατικός για τα θέματα αυτά. Το βασικό ερώτημα παραμένει όχι η ίδια η οδηγία, αλλά το πώς θα την εφαρμόσουμε από την οδηγία και αυτό προϋποθέτει και την απλοποίησή της. Σας ευχαριστώ για την σαφήνεια των λόγων σας. Από την πλευρά της Κομισιόν <clears throat> υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να λάβει τον λόγο. Κανονίστε μεταξύ σα ποιο θέλει, άμα δεν μπορείτε να αποφασίσετε θα δώσω λόγο στον εισηγητή. Ναι, θέλετε παρόλα αυτά να λάβετε τον λόγο. Παρακαλώ. Μιλάω εκ μέρους της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και εγώ θα ήθελα απλώ να πω ότι όλες οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερως χρήσιμες για μας και αντιλαμβανόμαστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχει επισημάνει η κυρία Ρούλε μόλις τώρα. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αποτέλεσμα της ε, ακρόασης τη Δετάρτη και κυρίως το αποτέλεσμα της έκθεσης και μπορώ να σας πω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εξεύρει μια καλύτερη προσέγγιση προκειμένου να υπάρχουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και να μπορέσουμε να τις ε, έχουμε όλες ε, συγκεντρωμένες σε έναν ιστότοπο ώστε κάποιος από κάποια τοπική αρχή να έχει πρόσβαση σε ένα συντονισμένο σύνολο κανόνων ψάχνοντας ε, λίγο πολύ μια μέρα στο διαδίκτυο τι δυνατότητες του δίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Um <laughs> Μερικές φορές φτάνει μια μέρα για να δει κανεί όλες αυτές τις παραλλαγές. Ο κύριο Λάσα και να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρέπει να δουλέψουμε από κοινού έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να εφαρμοστούν αυτές οι νέες διατάξεις. Καταφέραμε να απλουστεύσουμε και να αποσαφηνίσουμε την νομοθεσία και Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό ε, έχουμε πλέον στο απλοστάσιό μας ένα πάρα πολύ ένα καλό ε, μέσο κατά της ε, κρίσης. Μόλις εμφανιστούν επιπλοκές, ξέρετε, θα υπάρξουν και περαιτέρω προβλήματα, ανεργίες κτλ. Γι' αυτό λοιπόν προς το δικό μας συμφέρον θα πρέπει οπωσδήποτε οι διαδικασίες αυτές να γίνουν απλές, σαφείς και διαφανής. Άκουσα προηγουμένως και τον ε, Ισπανό Υπουργό και ε, με ευχαρίστηση άκουσα ότι μία από τις προτεραιότητες του είναι η απλούστευση των νομικών πλαισίων και η αποσαφήνιση κάποιων ελέγχων, πράγμα επίσης πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις παρατηρήσεις σας και για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να κλείσω τη συνεδρίαση και σας πενθυμίζω ότι συνεχίζουμε στις 9 το πρωί αύριο. Μην ξεχάσετε ότι συνεχίζουμε, υπάρχει συνέχεια.